Καλησπέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εγώ ήμουν στην ώρα μου πάντως, αλλά ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε όλους να καταφθάσετε πριν ξεκινήσουμε. Σήμερα, για τους πολίτες της Ευρώπης, συζητούμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το μέλλον της Ευρώπης, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα οποία θέλουμε να υποφεληθούν από τα όσα πράττουμε σήμερα. Προσπάθεια στην οποία πρέπει όλοι μας να επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας. Κυρίες και κύριοι, Έχουμε ένα νέο όνομα για το πρόγραμμα που θα συζητήσουμε, το Yes Europe. Νεολαία, εκπαίδευση, αθλητισμός. Αυτό σημαίνει το ακρονίμιο. Το νέο όνομα θέλει λοιπόν Yes Europe Επ' αυτού ψηφίζουμε άλλωστε. Οι συναδελφοί μου είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Έχουμε σχέδιο έκθεσης με ήδη 235 τροπολογίες. Υπό ότι οι συνθήκες δεν επιτράπησε όλους τους συναδέλφους να τροποποιήσουν το σχέδιό μου. Κινηθήκαμε με βάση το κείμενο της Κομισιόν, επί το οποίο υποβλήθηκαν 606 τροπολογίες, οι οποίες όμως εν μέρει καλύπτονται από τα δικά μου σχόλια, στην δική μου έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, αριθμός τροπολογιών δεν θα είναι δυνατόν ληφθούν πλήρω υπόψη. Αλλιώς θα γυρίσουμε πίσω από την αρχή. Η Ήτρα έχει υποβάλει 69 τροπολογίες, έχουμε 60 από την Επιτροπή Προπολογισμών, μια άλλη Επιτροπή 109. Λοιπόν, μιλάμε για πάνω από χίλιε τροπολογίε συνολικώ. Είναι αδύνατον να αποκτήσει κανεί σαφή εικόνα όλων αυτών. Α προσπαθήσουμε όμω να ομαδοποιήσουμε κάπως τη δουλειά μα και να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα κεφάλαιο για την νεολαία, για του νέου το οποίο δεν προϋπήρχε. Πρόκειται για ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού, όπως είπα ξεχωριστό κεφάλαιο, ξεχωριστός τίτλος. Το όνομα βεβαίως έχει αλλάξει, όπως σας είπα. Ξέρετε, το Κομινίου, στο Γκρουντβιχ, το Λεωνάρντο είναι άλλες πρωτοβουλίες στον χώρο της εκπαίδευσης που θα συμπεριληφθούν φυσικά υπό τον τίτλο εκπαίδευση. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, συμφωνήσαμε με βάση τις ε, υποβληθήσεις τροπολογίες να ξαναδούμε το πόσο για την εκπαίδευση και να κάνουμε κάτι ώστε να προβληθεί η δουλειά μας και τα προγράμματα τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Η Κομισιόν έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά τη. Στο κείμενο λέμε επίσης τι θεωρούμε ότι πρέπει να πράξει η Κομισιόν. Η Κομισιόν παρακαλώ με διορθώσει αν έχει την καλοσύνη. Έχει κάποια πρόταση ως προς την ακολουθητέα διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί δεν, αυτό σίγουρα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν. Επίσης, καλούμε τα θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία Ζαμονέ. Σχολιάζουμε και τις λεπτομέρειες. Για τα περισσότερα πάντως έχουμε συμφωνήσει. Να αναφερθώ λοιπόν τώρα στα εκρεμή επιμαχαζητήματα, αν μου επιτρέπετε. Ένα βασικό ζήτημα στο οποίο οι απόψει διήστανται και αυτό προκύπτει και από τις τροπολογίες αλλά και από όσο ένα γνώμη εκτός Κομισιόν είναι το θέμα της, ε, του μηχανισμού εγγύηση των δανείων για μάστερ. Αυτό με τους ε, σκιώδει εισηγητές και με την Κομισιόν το συζήτησαμε δις. Εγώ φίλο εξ να σας πω ότι είμαι υπέρ αυτής της δυνατότητας, υπέρ του μηχανισμού. Κανέναν δεν υποχρεώνουμε να λάβει αυτό το δάνειο, αλλά θα υπάρχει σίγουρα δυνατότητα. Πρόκειται για σημαντικό μηχανισμό, ο οποίο θα διευκολύνει του φοιτητέ που κάνουν το μάστερ του στο εξωτερικό. Είτε πρόκειται για μονοετέ είτε για διαιτέ μάστερ. Επίση, θα διευκολύνει ανθρώπου που ενδεχομένω δίσταζαν να πάρουν δάνειο. Υπάρχουν κάποιοι που τάσσονται κατά του μηχανισμού, ζητούσαν επιπλέον εγγύησει συγκεκριμένα. Εν προκειμένου η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένω να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ο μηχανισμό έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε κοινωνικά αιτήματα, να είμαστε πιο ευαίσθητοι και να μα πείτε βεβαίω και πού καλύπτεται το θέμα αυτό στην πρότασή σα. Οι διδακτορικοί φοιτητέ είναι επίση μια άλλη σημαντική ομάδα. Πρόκειται για μια ομάδα στόχο όσον αφορά την κινητικότητα και το λέμε αυτό στην έκθεση. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αναφερθούν ξεχωριστά. Είναι φοιτητέ είτε προπτυχιακοί φοιτητέ, είτε στο στάδιο του μάστερ του διδακτορικού, όλοι είναι φοιτητέ. Πάντω, ειδικά για τα μάστερ και τα δάνεια, φοβούμαι ότι τα δάνεια αυτά μπορούν να προσφερθούν σε φοιτητέ σε επίπεδο μάστερ, αλλά θα ήταν υπερβολικά δαπανηρό να δίνονται και στους διδακτορικούς φοιτητές. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα έχει να πει δύο πράγματα για όλα αυτά. Στο πρόγραμμα, στον ορίζοντα μάλλον 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένω να μας διευκρινίσει, επαναλαμβάνω, το πώς βλέπει όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τον στόχο του προγράμματος συνολικός, οι επιμέρους στόχοι για επιμέρους συγκεκριμένες ε, κατηγορίες ε, προκάλεσαν την υποβολή πολλών τροπολογιών. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε είναι τα υπερπόντια διαμερίσματα και χώρες, ακριβώς επειδή έχουν τις δημορφίες τους. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, ε, δεν χρειάζεται να το δούμε ως πρόβλημα, οι χώρε αυτή τη ομάδας, τα υπερπόντια διαμερίσματα, είναι τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, για παράδειγμα, είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αναφερθούν ονομαστικώ. Καλύπτονται εκ των πραγμάτων από την πρότασή μα. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή αναφορά. Επίση το Erasmus Mundus. Είναι ένα πασίνωστο πρόγραμμα και θα είναι ένα στο πρόγραμμα. Συμφωνούμε ότι αυτό το όνομα θα χρησιμοποιούμε και στο μέλλον. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, το ράσμους μούντους θα αναφερθεί στο πρόγραμμα. Πρόκειται για πρόγραμμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια πολύ γνωστή επωνυμία, αν θέλετε. Κατά τα άλλα, κάποιοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την διεθνή διάσταση του προγράμματος όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση. Όσον αφορά δηλαδή, δηλαδή την κινητικότητα για τους φοιτητές της τεχνικής εκπαίδευσης της, στο στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Εγώ πιστεύω ότι η κινητικότητα σε αυτόν τον τομέα και μάλιστα σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Είναι κάτι εκτός της εντολής μας και δεν έχουμε και τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσθέσει ένα κεφάλαιο για την κινητικότητα και ένα άλλο για την διεθνή συνεργασία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρω ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την συνεργασία μας με τρίτες χώρες, τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Όσον αφορά όμως την κινητικότητα, νομίζω ότι αυτά εκφεύγουν τις εντολής μας. Επίσης, στο κεφάλαιο αθλητισμός, και εδώ είχαμε πολλές προτάσεις, εν γέννη μια συντριπτική πλειονότητα τάστε υπέρ τη ανάπτυξης των τομέα και κατά των διακρίσεων. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και την εθελοντική εργασία για να ενισχυθούν οι δεσμοί με τον χώρο του αθλητισμού. Θα προσπαθήσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες να τις αποτυπώσουμε στην έκθεση. Ένας άλλος τομέας, στον οποίο λάβαμε πολλές τροπολογίες, ένα άλλο επίμαχο ζήτημα επί του οποίου θα προσπαθήσω να καταλήξω σε συμβασμό, είναι η σύνδεση της πόλης με τον αθλητισμό. Αλλά αυτό το είδαμε, λέει η μιλήτρια. Με συγχωρείτε, γιατί έχω εδώ όλα τα χαρτιά μαζεμένα μπροστά μου. Αυτά, μάλλον. Το γεγονό είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές τροπολογίες, το, τα δάνεια για το μάστερ, τον αθλητισμό, έχουμε το θέμα του προπολογισμού βεβαίω. δεν το είπα, έπρεπε. Τρία λοιπόν τα βασικά ζητήματα Επί αυτών των ε, τριών ζητημάτων ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Γιατί είναι καθόδη ζητήματα όντως. Ελπίζω να συμφωνείτε με την πρότασή μου να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις τροπολογίες σε συμβαστικές. Ο διάλογος ε, στο Κοινοβούλιο δεν εξαιρετικά επικοδομητικό. Νομίζω ότι σπάνια βλέπουμε τόση εργασία. Ε, στις 22 ε, Νοεμβρίου ψηφίζουμε. Μέχρι τώρα θα τα πούμε με τους σκιώδεις. Έχουμε πολλές ευκαιρίες. Και ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα υποστηρίξει σύσσωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιόντε Κουρέλ θα είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να παραδεχθώ ότι θα είμαι πολύ φιλική προς την Κομισιόν. Ξεκίνησε επιθετικά, πολλά δεν έγιναν στην αρχή, αλλά τώρα πια πραγματικά οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια, για τη βοήθειά σας, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ελπίζω ότι μαζί θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έχουμε έναν ε, κοινό φίλο ή εχθρό, <laughs> όπω το πάρετε, στο Συμβούλιο, το λεφτό προς την Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα τι έχουμε μπροστά μας. Ε, έχουμε μακρύ κατάλογο μιλητών. Μαρίτα Σάντσες Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενοι στην πρόταση της ε, Κομισιόν και τον τίτλο που είχε δώσει η Κομισιόν σε αυτό το φάκελο, το Εράσμους για όλους, ε, σκοπός ήταν να μην ε, ξεχάσουμε κανέναν και να... Και αυτή η διάταξη που επιτρέπει την κινητικότητα να είναι προσπελάσιμη στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων. Γι' αυτό το λόγο ήταν τόσο πολλοί άριθμες τροπολογίες επί του θέματος. Αληθεύει ότι είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με τα άτομα αποδέκτες ε, αυτού του μηχανισμού. Υπάρχει μια διευκρίνηση. Τι πώς εννοούμε τον όρο σπουδαστής, φοιτητής, καλύπτει ευρέως ε, όσους ε, παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε για τον ορισμό αυτού του όρου, διότι σε κάθε χώρα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες ατόμων ε, όσον αφορά μάλιστα την επαγγελματική κατάρτιση. Τέθηκε το ζήτημα ότι αυτός ο μηχανισμός κινητικότητας θα ανοιχτεί σε όσους ε, ε, ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση ενώ σε κάποιες χώρες ε, ανοίξει συγκεκριμένες κατηγορίες και σχετίζεται με συγκεκριμένα πανεπιστήμια ενώ σε άλλα κράτη σχετίζεται με ιδρύματα ανεξάρτητα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επιθυμούσα λοιπόν αυτοί οι μηχανισμοί κινητικότητας να ανοίξουν για φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο βρίσκει συνένεση και δεδομένου βέβαια του, των, των δημοσιονομικών μας περιορισμών θα προσπαθήσουμε να σε στηρίξουμε όλοι ώστε να επιτύχουμε έναν επαρκή προπολογισμό ώστε να καλύψουμε τις φιλοδοξίες μας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε όσου ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση από αυτό το μηχανισμό κινητικότητα. Το δεύτερο σημείο που φαίνεται ενδιαφέρον είναι αυτό το σύστημα των δανείων προς τους φοιτητέ. Θα επιθυμούσα να μην αντικαταστήσει τις υποτροφίες που απευθύνονται σε άλλο κοινό. Να μην αντικαταστήσει λοιπόν αυτές τις υποτροφίες διότι εκεί απομακρυνόμαστε υπερβολικά από το στόχο μας. Το τρίτο θέμα που με ανησυχεί νομίζω βρίσκεται στο άρθρο 7 όσοι αναζητούν εργασία επειδή έχουν μόλις βγει από το πανεπιστήμιο και νομίζω στη συμβιβαστική πρόταση προτάθηκε η περίοδος που δίνει δικαίωμα κινητικότητας να περιοριστεί σε 10 μήνες, σε 12 μήνες, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις χρηματοδοτήσεις που θα θέλαμε. Είναι σημαντικό οι νέοι που βρίσκονται σε αυτή τη ε, θέση αναζήτησης εργασίας και που μπορούν να ε, έχουν κάποια, να λάβουν κάποια ε, υποτροφία ε, να μπορέσουν να ενταχθούν στο χώρο εργασίας. Και το τελευταίο θέμα που θεωρώ σημαντικό είναι ο αθλητισμός. Πρόκειται για μια νέα αρμοδιότητα και προσπαθούμε να ορίσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να υποστηρίξει τον αθλητισμό Ε, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, ανθρώπους νεότερης ηλικία και θα πρέπει να καταφέρουμε στον τομέα του αθλητισμού να ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους από τις χαμηλότερες δυνατές ηλικίε ώστε να αποτελεί ε, αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής ο αθλητισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Προσπαθώ να τον αντικαταστήσω τον κύριο και του εύχομαι το καλύτερο αποτέλεσμα αυτή την Κυριακή. Ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία που υπέβαλαν πολλοί συνάδελφοι αυτής της Επιτροπής σε σχέση με το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα διεθνές πανεπιστήμιο, έργο ενός ευρωπαϊκού έργου της ε, Ένωση για τη Μεσόγειο που αποτελεί κομμάτι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Είναι ουσιαστικά το μοναδικό άμεσο μέσο αυτής της πολιτικής και υποστηρίχθηκε ευρέω από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ε, και ειδικότερα από τον πρόεδρο της Κομισιόν του κ. Μπαρόσο αλλά και άλλους πολιτικούς. Σκοπός του Πανεπιστημίου αυτού είναι η συνεργασία στο Ευρωμεσογειακή Λεκάνη, στη Λεκάνη της Μεσογείου ουσιαστικά, τον πρώτο χρόνο ίδρυσής του, στα πρώτα του βήματα, το πανεπιστήμιο αυτό εστιάστηκε στην προβολή του και την καθιέρωση ενός ευρώς δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά γιγάντιο, διότι ήδη σήμερα συνεργαστεί με 206 ιδρύματα ερευνητικά από 42 χώρες. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ε, στελεχών, ε, υπάρχουν κάποιες νέες θέσεις στο Πανεπιστήμιο και ε, όλο αυτό το προσωπικό έχει πολύ φιλοδοξούς στόχους. Μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο διοργανώνει συνέδρια, καλοκαιρινά μαθήματα, επαγγελματικά μαθήματα και τώρα η ηγεσία του Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να αποτελέσει το Πανεπιστήμιο αυτό ένα λειτουργικό και καλά παγιωμένο Πανεπιστήμιο. Ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, φυσικά χρειάζεται υποστήριξη όχι μόνο ηθική αλλά και οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε αυτό το πρόγραμμα που αφορά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσα είπαμε ήταν οι στόχοι μας και οι πολιτικές μας και οι στόχοι μας αυτοί θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κώστα. Η κυρία είναι πρώτη. Η κυρία Σφίνμπορν είναι πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ την Έμα Μακλάκιν από την πολιτική ομάδα ECR. Δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ λόγω υποχρεώσεων στην εκλογική τη περιφέρεια. Όμω υπέβαλε διάφορε τροπολογίε. Θα ήθελα να τονίσω ορισμένε από αυτέ. Όσον αφορά τον αθλητισμό, η ομάδα ECR πιστεύει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στον αθλητισμό στη βάση. Υποστηρίζουμε την προαγωγή τοπικών πρωτοβουλειών από την τοπική κοινωνία. Οι οργανώσεις βάσης, τοπικές αθλητικές ενώσεις πρέπει να αποτελέσουν, αν θέλετε, τη ρεχοκοκαλιά αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτές θα παίξουν τον βασικό ρόλο σε μια, για μια περιεκτική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο, δεν πρέπει να είναι απαραίτητο αυτές να είναι διεθνικές, όπως έχει γραφτεί σε κάποιο σημείο. Η προαγωγή επίσης του εθελοντισμού στον αθλητισμό είναι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου με αφορμή του Ολυμπιακούς ε, νομίζω το απέδειξε πόσο, μπορούν, πόσο θετικά μπορούμε να επηρεάσουμε τους συμμετέχοντες. Επίσης, ε, όσον αφορά την διαγραφή στην χρηματοδότηση. Οι τοπικέ πρωτοβουλίε δεν είναι δυνατόν να έχουν εμπορικά έσοδα, όπως υπονοεί το κείμενο. Θεωρώ ότι πρέπει να διαγράψουμε εδώ ένα κομμάτι του κειμένου για να μην υπάρχει μια αντίφαση με την ανάγκη ακριβώ χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν οι συμπράξει με τρίτου είναι ένα πολύ σημαντικό περιουσικό στοιχείο, αν θέλετε, και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Θέλουμε να περιληφθεί αυτή η δυνατότητα εξασφάλιση εμπορικών εισόδων. Κύριε Μακλάχλιν, επίση, θέλει μείωση του προβλησμού Ζωαμονέ. Ο προβλησμό για τον πολιτισμό θα έπρεπε να εστιάζεται στην προσθεμένη αξία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να ξοδέψουμε περισσότερα στο συγκεκριμένο ε, θέμα από ότι για ολόκληρο το κομμάτι που αφορά τον αθλητισμό. θα μπορούσαμε ε, νομίζω να βρούμε προσθεμένη αξία αλλού. Όσον αφορά επίση τι εγγυήσει των δανείων και το πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα στην πράξη, πιστεύουμε ότι ε, ενδεχομένω εδώ επεκτείνουμε με επικίνδυνο τρόπο την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι για να ε, αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά η προσπάθεια θα είναι δύσκολη. Η εμπειρία μας με τα δάνεια για φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι είναι δύσκολο τα δάνεια αυτά να αποπληρωθούν από τη στιγμή που φεύγουν από τη χώρα στην οποία σπούδασαν και όπου έλαβαν το δάνειο για να ζήσουν σε άλλη κοινωτική χώρα ή αλλού. Συνεπώς, μια, ένας τέτοιος μηχανισμός θα επιφέρει, θα δημιουργήσει επιπλέον βάρος το οποίο θα φέρουμε μακροπρόθεσμα. Τέλος, όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες της CCR δεν έχουν ίσως ακόμη συμπεριληφθεί στην προσπάθεια αυτή, οπότε περιμένουμε τα σχόλια της ε, Πρόεδρου. Σας ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι. Λεκεγκάρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια και βρισκόμαστε μέσα στις διαπραγματεύσεις, καλό είναι νομίζω να πούμε δύο λόγια για αυτές τις διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα. Θα έλεγα ότι μπορώ να πω ότι τα πράγματα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Νομίζω είχαμε καλές συναντήσεις, θετικές. Κάποια λίγα σχόλια θέλω να προσθέσω για τις κυριότερες ανησυχίες ως, ως μελήματα μέχρι σήμερα. Δεν είναι μυστικό για μας από την Άλντε. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει ισορροπία μεταξύ απλούστευσης και σαφήνειας. Μια και τώρα που ελπίζουμε σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής να έχουμε θετική έκβαση. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ απλούστευσης και όπως ελπίζουμε και την αύξηση των κονδυλίων από πλευράς προϋπολογισμού. Γι' αυτό είναι θετικό το ότι εργαζόμαστε σε μια πιο απλουστευμένη διατύπωση Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι να τα πετύχουμε. Η Άλντε έχει τροπολογίες με αυτή την προσέγγιση υπόψη για τα άρθρα 5, 7, 8 και 10. Ελπίζω ότι θα έχουμε καλά θετικά αποτελέσματα στο τέλος τέλος για τις διαπραγματεύσεις που επικίνδυνε για αυτά τα θέματα. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το άρθρο 13, προτείναμε κάποια ποσά εμείς ανατομής. Κατά 76% προσθήκη, δηλαδή προς 35% για την ανώτατη εκπαίδευση, 18% για τη σχολική εκπαίδευση, 5% ε, όσον αφορά τις ε, ειδικέ δράσεις ε, πρόσθετης αξίας. Σε σχέση με την κίνηση για την νομική βάση, συμφωνώ ότι αυτό ήταν το σωστό που έπρεπε να γίνει. Και νομίζω ότι Προς αυτή την προσέγγιση κινούμαστε. Πρέπει να συμφωνήσουμε τώρα για τα ποσά τελικά και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σε σχέση με το μέσο διευκόλυνσης για τα δάνεια, για τις ε, πιστώσεις, είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε αλλάξει τη θέση μας και έχουμε μετακινηθεί. Μπορούμε να δούμε σε σχέση με το Συμβούλιο όπου τα κράτη-μέλη είναι διχασμένα εκεί και για αυτό το θέμα. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν διαφορετική χρήση αυτού του μέσου, αυτής της διευκόλυνσης για να το πω με απλά λόγια, θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα από κάποια κράτη σε σχέση με άλλα. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό έχουμε κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τα σκανδιναβικά κράτη για αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δούμε την κατάσταση που θα πρέπει να επιτύχουμε να είναι αποδεκτή για όλους. Δεν βρήκαμε ακόμα την χρυσή πορεία και έχουμε και το θέμα του κανονισμού και είναι δύσκολο να κάνει κανείς λόγο για εθελοντική, εθελούσια συμμετοχή για τα κράτη-μέλη. Πρέπει όμως να ξανασκεφθούμε τα πράγματα άλλη μια φορά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε τη δική μας, να υπάρχει δική μας υποστήριξη. Δεν είναι σωστά τα πράγματα όπως προτάθηκαν και όπως έχουν τώρα. Θα πρότεινα να ξαναδούμε ακόμα μια φορά τα πράγματα, να δούμε μήπως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον Erasmus Mundus, τον έρασμο για όλους. Νομίζω έχει δίκιο η Πρόεδρος. Ίσως θα έπρεπε τελικά να έχουμε κάποια αναφορά σε αυτό το πρόγραμμα. Συγκεκριμένη αναφορά. Πολλοί είναι οπαδοί και ένθερμοι οπαδοί του Εράσμου για όλους. Και μια και γίνεται η προσπάθεια σε σχέση με τους τίτλους, ονομασίες, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το Εράσμος Mundus. Τουλάχιστον να υπάρχει ένα ακόμα Εράσμος που θα μπορεί να, να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτά είναι τα σχόλια από πλευράς μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Έχουμε προσεγγίσει, θα έλεγα, πολύ τις θέσεις μας. Εξαιρετικό. Κύριος Καβαντά, παρακαλώ. Ζαν Μαρή Καβαντά, έχετε τον λόγο εντυπωσιάστηκα από την καλή σας κίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια μικρή παρατήρηση. Ο συναδελφός κύριος Λάκεγκάρντ, όπως και εσείς, ε, έχει δίκιο. Χρειάζονται χρόνια για να δημιουργήσει κανείς μια δημοφιλή μάρκα. Θα ήταν ανόητο λοιπόν να την πατάξουμε σκουπίδια. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω, κυρίες και κύριοι, να μην χαλάσουμε κάτι που ήδη λειτουργεί καλά. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και βασίζομαι σε όσα είπε η κυρία Πρόεδρος αλλά αυτό που ευθύνεται κιόλα και σε ολόκληρη την Επιτροπή θα ήθελα κάπου να αναφέρεται έστω και σε ένα προήμιο ή τουλάχιστον σε μια αιτιολογική σκέψη κάποια διατύπωση που να εκφράσει την ακολουθή ιδέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκε από ιδρυτικές πράξεις το 1950 σε το 1900, η ΕΟΚ, αργότερα η κοινή γεωργική πολιτική και τέλος το ευρώ. Και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων που κανείς δεν θυμάται με ακρίβεια. Όσον αφορά το Εράσμους, δεν χρειάστηκε πολύ καιρό ώστε αυτό το σήμα να εκτυπωθεί και να αναρτάται σε ε, όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους και Ήδη γυρίζεται η τρίτη ταινία, το Ισπανικό Πανδοχείο αριθμό 3 ε, γαλλικής παραγωγής που βασίζεται στο Εράσμους. Θα ήθελα να σημειωθεί ότι αυτή η τεράστια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν οδήγησε ποτέ σε καμία αντίφαση, αντίθετα με την κοινή αγορά, το να είναι ανεπαρκής. 3% των φοιτητών σε μία ήπειρο που έπρεπε να χρησιμοποιεί τους φοιτητές ως βασικό θεμέλιο λίθο θα έπρεπε να υποστηρίζουμε την ιδέα ότι αυτή η τεράστια επιτυχία είναι ανεπαρκής και χρειάζεται να αφιερώσουμε μέσα για να, για να τη διευρύνουμε. Πολύ σημαντικά είναι έγκλημα το να βλέπουμε μια τέτοια υπόθεση που λειτουργεί, που αποτελεί μια καταπληκτική σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, ισχυρό σημείο της Ευρώπης. Ναι, συζητάμε φυσικά τους προπολογισμού και είναι φυσιολογικό σε περίοδους κρίσης. Αλλά εγώ, εγώ μιλάω για τα 25 χρόνια που μας χωρίζουν από το 1987, όπου σήμερα θα έπρεπε να αφιερώνουμε υποτροφίες και να χρηματοδοτούμε τους νέους για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί αυτή είναι η βάση του ό,τι γίνεται, του ό,τι καλού γίνεται στην Ευρώπη μεταξύ των πολιτών. Σας ε, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα βρείτε με το ταλέντο σας μια καλή διατύπωση ή διαφορετικά θα σας κάνω και εγώ μια πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία και δυστυχώς αρκετά ακόμη περιορισμένη παρά την τεράστια φήμη της. Ευχαριστώ. Je... Je vais le... Θα το σκεφτώ. Είχαμε ωστόσο μια προθεσμία για τις τροπολογίες. Αν πρόκειται λοιπόν να υποβάλλετε τροπολογία, κάντε τη σύντομη και προφορική. Να, να τη συζητήσουμε κατά την ψηφοφορία, αλλά κάντε την όσο το δυνατόν ταχύτερα, ώστε να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα είναι τρεις σειρές το πολύ, τρεις γραμμές το πολύ. Ναι, αλλά η προθεσμία ισχύει είτε για τρεις είτε για πέντε γραμμές. Ε. Διότι μου έκανε έκπληξη που δεν βρήκα κάτι τέτοιο εκεί μέσα. Συμφωνώ, λέει η Πρόεδρος. Θα δράσουμε. Θα επιληφθούμε του θέματος. Και τώρα η κυρία Ναβενάλογα. Ďakujem Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω πράγματα που ανέφεραν ήδη οι συναδελφοί. Δεν είναι αυτή η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το Εράσμους εδώ στην Επιτροπή μας. Η συνεργασία μας ε, υπήρξε ε, ιδιαίτερα διαφωτιστική και χαίρομαι που καταφέρα να συμμετέχω και εγώ και να προσφέρω στις, δεν συνεισφέρω στις συζητήσεις. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τα βασικά σημεία του προγράμματος, συμμετοχή, κινητικότητα. Θα πρέπει να εστιαστούμε και στην επέκταση αυτής, ε, αυτού του μηχανισμού, αυτής της υπηρεσίας σε όλους τους πολίτες. Πολλοί συνάδελφοι προσπαθούν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή του προγράμματος ώστε να συμπεριλάβει και τους ενέργους. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας ε, εάν ε, επεκτείνουμε υπερβολικά το Εράσμους. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να μην έχουμε αρκετά κονδύλια για τους νέους ώστε να συμπεριληφθούν για παράδειγμα οι αθλητικές δραστηριότητες. Φυσικά με ικανοποιεί που βλέπω τόσες πολλές τροπολογίες, έχουμε κάποιες εξαιρετικές συμβαστικές τροπολογίες. Είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρουμε να ε, τις διεκπαιρεώσουμε και να καταλήξουμε σε επιτυχείς, σε επιτυχείς συμβιβασμούς. Καταφέραμε να επιτύχουμε κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας τη γενική ομολογία δεν θα πρέπει να αποφασίζουν μόνο τα θεσμικά όργανα, αλλά και όσοι επηρεάζονται πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παρατηρώ ότι αυτό έχει προταθεί και όσον αφορά το σύστημα δανείων. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το ζήτημα. Η ομάδα μας έχει καταλήξει σε μια πρόταση την οποία έχει υποβάλει. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές από μας έχουν ληφθεί υπόψη. Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει κοινή τροπολογία. Ο κ. Λέκεγκαρντ δεν ήταν παρόν σήμερα για τη συνεδρίασή μας. Συναντηθήκαμε με την Κομισιόν. η οποία σαφώς εξήγησε την πλέον πρόσφατη πρόταση. Η Κομισιόν προτείνει ένα κείμενο που πλησιάζει όλο και περισσότερο την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και για αυτό το θέμα θα πρέπει να προβληματιστούμε. Η σημερινή μας συνεδρία ήταν πολύ καλή, η σημερινή μας συνάντηση και ευελπιστώ ότι αύριο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα και να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο για τον προϋπολογισμό τώρα ακόμα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά θα πάρουμε τα κονδύλια αυτά τα οποία επιθυμούμε αν υπάρχει εκπρόσωπος της Προεδρίας απόψε θα χαιρόμουν αν μπορούσε να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε από κοινού όλοι. Σε ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω γι' αυτό το χαρτοφυλάκιο, όσους όσους εργάστηκαν σε αυτό. Δύσκολη η συνένεση, αλλά την πετύχαμε, τα καταφέραμε. Με την συγγήτρια συμφωνώ για τα θέματα για τον προϋπολογισμό. Ή μάλλον αυτό είναι ένα ερώτημα περισσότερο, ένα ζήτημα το οποίο απομένει. Αφορά τους υπουργούς μας, εκείνους που μέχρι σήμερα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα αν για το Yes Europe σήμερα μπορούν να πούν κατεκτήμηση είναι έστω κιόλας πώς θα έχουν τα πράγματα συνολικά με τον προϋπολογισμό, τι θα γίνει με τα κονδύλια συνολικά και με τα επιμέρους προγράμματα ατομιακά, επιμέρους εξειδικευμένα. Θα ήταν σημαντικό να τα γνωρίζαμε αυτά. Πώς τα βλέπετε εσείς κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς υπάρχουν εκεί για παράδειγμα τουλάχιστον κάποιες ποσοστώσεις για κονδύλια για τα επιμέρους αυτά σημεία ή θα αλλάξει κάτι, υπάρχει κάποια μεταβολή. Πώς τα βλέπετε. Θα μπορούσαμε ίσως και τουλάχιστον να έχουμε περισσότερα κατελάχιστον κονδύλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπέναρα τους παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, υπογραμμίζω ότι συζητήσαμε, συνηθήκαμε κατά επανάληψη. Χάρη σε αυτό κατορθώσαμε να διαμορφώσουμε θέση στην έκθεση για το αίρεσμο. Στέκομαι σε αυτά όσα είπε ο κ. Καβαντά. Το αίρεσμο είναι γνωστό, πασίγνωστο. Όσον αφορά τον προπολισμό, ο κ. Λαμασούρ είπε ότι υπάρχει κίνδυνος της χρηματοδότησης του αίρεσμο. Αυτό θα δείξει πάρα πολλούς και θα είναι τρομερό. Είναι τόσο γνωστό το αίρεσμο. Πολλοί περιμένουν πολλά από το αίρεσμο. Το επιχείρημά μα είναι ότι το Yes Europe είναι και πάλι αγγλόφωνο σύνθημα. Θέλουμε για λόγους πολυφωνίας και μόνο κάθε φορά που προκρίνουμε έναν τίτλο, ένα σύμβολο, να είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στι άλλε γλώσσε. Ενώ εδώ χρησιμοποιούμε αναγκαστικά τα αγγλικά. Υποστηρίζω λοιπόν την τροπολογία του κ. Καβεντά. Έρασμος για όλους. Όντως δεν είναι... ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου αρχικώς. μικρόφωνο, δεν ακούστηκε η πρόεδρο. Θέλεις να προσθέσουμε κάτι στο προήμιο. Ναι. Θυμίζω ότι είπα προηγουμένως. Ναι, φυσικά είπα έρασμος για όλους. Το είπα, το είπα στην αρχή. Είπα, επαναλαμβάνω, ότι το έρασμος είναι μια γνωστή επωνυμία και να την κρατήσουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Συνεχίστε παρακαλώ. Συνεχίζω. Όσον αφορά το θέμα των εγγύσεων των δανείων, σημαντικό. Τα είπαμε με την Κομισιόν κατά επανάληψη, εγώ πιστεύω ότι ο στόχος των εγκυμένων δανείων είναι περισσότεροι φοιτητέ να μπορέσουν να κάνουν ένα μάστερ στο πλαίσιο της κινητικότητας. Αν συμφωνούμε με τον στόχο, τότε με βάση κοινωνικά κριτήρια ας πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Η Κομισιόν φαντάζομαι θα μας προτείνει κάτι για να έχουμε μια βάση για τη συζήτηση. Και κάτι άλλο. Προϋποθέσεις χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Σημασία έχει να μην επιλέγουν συγκεκριμένες σχολές τράπεζες. Όλα να κρίνονται επί ίσης όρης. Ίση πρόσβαση. Τώρα, πιστεύω ότι από αυτού θα κατορθώσουμε να συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω αν είμαι αισιοδόξη. Και τέλος, για την ε, διεθνή συνεργασία Εράσμος Μοντούς. Ψηφίσαμε, θυμίζω, με συντριπτική πλειονότητα, μια γραπτή δήλωση για το Έρασμος Euromed, το ευρωμεσογειακό Έρασμος, εδώ και μήνες. Το Έρασμος Μόντους καλύπτει τον πλανήτη, αλλά θα μπορούσαμε στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας και λόγω της συνεργασίας που έχουμε να κρατήσουμε και το Erasmus Euromed, κομμάτι δηλαδή του Erasmus Mundus. Πάντα παραλαμβάνω στο πλαίσιο της γειτονίας. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ζωής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τη Μεσόγειο, της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης θα λέω ότι πρέπει να κάνουμε και αυτό το βήμα προς ένα δίκτυο πανεπιστημίων, ίσως και ένα ευρωμεσογειακό ε, δίκτυο, το οποίο θα, μπορεί, θα μπορέσει να στηριχθεί στο Erasmus EuroMed. Ευχαριστώ. Τώρα εξαντλήθηκαν όλα τα ερωτήματα. Ωραία. Θα ήθελα ίδια να πω δύο λόγια και μετά δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως μπορεί να διορθώσει αν κάνω κανένα λάθος. Ξεκινώ από την αρχή γιατί η Μαρή Τερές πρέπει να φύγει. Μαρή Τερές δεν πιστεύω ότι με κατάλαβες σωστά οι επαγγελματικές σχολές συμπεριλαμβάνονται και η κινητικότητα των μαθητών των επαγγελματικών σχολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνεται και αυτή. Οι άλλες ε, τροπολογίες ε, είναι διεθνούς χαρακτήρα και δεν μπορούμε να ε, χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δράσεις. Κινητικότητα για τους, τους μαθητές αυτών των σχολών, αυτό είχα πει. Δεν έχουμε τα χρήματα για να καλυφθούν όλες αυτές οι δράσεις. Οι επαγγελματικές σχολές είναι étudiants, είναι φοιτητές αυτοί και θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο υπό το πλαίσιο του παλαιού προγράμματος Λεωνάρντο. Μετά έχουμε το θέμα με τους 12 μήνες για τη διάρκεια. Από πλευρά τη κυρία Νενταλόβα αναφέρθηκε. Έχουμε μια δυνατότητα να καλύψουμε μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και γι' αυτό περισσότερο επικεντρωθήκαμε στην κατάρτιση και εκπαίδευση και όχι τόσο πολύ σε ε, άλλο πλαίσιο. Αλλά ίσως αυτούς τους 12 μήνες για τους οποίους γίνεται τώρα λόγος, για εκείνους που θέλουν να βρουν τέτοια απασχόληση, μπορούμε να διευρύνουμε. Η Επιτροπή μπορεί τους 12 να τους κάνει 14 ή 15 μήνες, να επεκτείνει την διάρκεια. Και αυτό είναι ένα θέμα που συνεπάγεται και χρηματοδοτικούς κινδύνους. Το θέμα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είχαμε ένα πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε από τα έξι θεσμικά όργανα και τέσσερα διέγραψε, δύο διατήρησε. Είπαμε είναι άδικο αυτό. Ή όλα θα διαγραφούν ή όλα θα παραμείνουν. Και αυτό έκανε το Συμβούλιο και παρέμειναν όλα. Αλλά δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε καινούρια, να εντάξουμε και άλλα θεσμικά όργανα, άλλα ιδρύματα. Και μόνο και μόνο η ιδέα αυτού του ιδρύματος είναι εξαιρετική ιδέα αλλά εγώ σε σχέση με τα Ιταλικά πανεπιστήμια τα γνωρίζω τα πράγματα πως έχουν και μπορώ να σας πω ότι τα Ιταλικά πανεπιστήμια εργάζονται πολύ στενά, στενά με τα μεσογειακά πανεπιστήμια. Το κάνουν ήδη. Δεν είναι ότι πρέπει να επινοήσουμε τον τροχό εξ αρχής. Γίνεται αυτό ήδη. Ουσιαστικά αυτή η ιδέα, στο πω έτσι, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργεί Πήγα στη Μπολόνια και το κάνουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 15 χρόνια. Αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Η ιδέα είναι καλή, αλλά εγώ η ίδια μια τέτοια τροπολογία δυστυχώς δεν μπορώ να την υποστηρίξω, διότι θα έπρεπε να υποστηρίξω και άλλες τροπολογίες με το ίδιο σκεπτικό και δεν έχουμε τα χρήματα για να ξεπεράσουμε τα έξι ιδρύματα. Είμαι με ανοιχτό πνεύμα ε, επικοδομητικής συνεργασίας, αλλά από πλευράς εισηγήτριας πρέπει να πω την άποψή μου και αυτό ίσως δεν ταιριάζει σε όλους σε εσά τώρα, εξ ονόματος, της κυρία, ε, ε, Μακλάκιν, για τα αθλήματα, κάποιες από τις προτάσεις σας εντάχθηκαν για τον αθλητισμό. Πολλές τροπολογίες κατατέθηκαν. Έχουμε, δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά ώστε να έχουμε μια χειροπιαστή πρόταση που να μπορεί να λειτουργήσει. Αύριο το πρωί θα έχουμε το, τη δυνατότητα να αποσταλεί αυτό στο Προεδρείο. Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι σημαντική βέβαια δεν μπορούμε, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το σημείο κοντά στο Λονδίνο, να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Εδώ πρόκειται για την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τοπικές πρωτοβουλίες που δεν έχουν καμιά σχέση με την ευρωπαϊκή διάθεση, διάσταση. Για αυτά τα θέματα είναι το Λονδίνο ή το Εδιμβούργο ή οι αρμόδιοι τοπικά στο κάθε κράτος υπεύθυνοι. Τώρα για τις απόψεις Μακλάρκιν ή με εσάς ε, κατανοώ τις ε, ιδέες σας και τις προτάσεις σας αλλά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι που δεν έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Όχι επειδή δεν είναι καλό αλλά επειδή δεν είναι δουλειά μας. Είναι δουλειά ή του Εδιμβούργου ή του Λονδίνου να υποστηρίξουν τέτοιες τοπικές πρωτοβουλίες. Μετά για το, τη διευκόλυνση για τα δάνεια για την αρμοδιότητα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω έτσι. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και χρηματοοικονομικά πιστοτικά ιδρύματα στα επιμέρους κράτη. Δεν το βλέπω έτσι, αλλά κατανοώ γιατί το λέτε και το προτείνετε. Κύριε Λόκεγκαντ, με τη διαφορά για το όφελος είναι δύσκολα τα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα, να γίνει κατανοητό είπαμε εντάξει δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί έχουμε ένα μέσο και οι Γερμανοί έχουν και οι Φινλανδοί και... αλλά πρόκειται για μια πρόσθετη ιστορία ως διάσταση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό που γίνεται φυσικά έχουμε πολλούς στη χώρα σας που για ένα δανέζικο π.χ. ή μια δανέζικη υποστήριξη αναφέρονται σε αυτήν και αυτοί χρησιμοποιούν γιατί είναι ίσως πιο ευνοϊκοί και γι' αυτό να μην ανταποκριθεί κανείς σε μια τέτοια ε, πρόταση γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να, ε, να ανταποκριθεί αλλά αν σκεφτούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο πόσοι φοιτητές ε, εράσμους υπάρχουν από εκεί. Όχι τόσοι όσοι σε σχέση με εκείνους που θέλουν να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί δεν το επιθυμούν. Δεν είναι δική μας δουλειά όμως να αναμειχθούμε και να το διευθετήσουμε. Βλέπετε το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται με εθελούσια εθελοντική βάση. Τα προγράμματά μας στοχεύουν σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κάθε αυτός πολίτης αν επιθυμεί να μπορεί να συμμετάσχει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αποκλείουμε. Δεν μπορεί λοιπόν κάτι να γίνεται εθελοντικά. Τώρα εθελοντικά κάποιο να παρετηθεί να πει εντάξει παρετούμε. Αν θέλει όμω να το αποκτήσει και δεν του το προσφέρουμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται με κανένα πρόγραμμα μια τέτοια εθελοντική, σε, με βάση, ούτε με το πρόγραμμα κομμένιους ούτε με το έρασμο. Δηλαδή τι να πούμε, δεν θα συμμετάσχουμε με το, στο πρόγραμμα ε, ο φοιτητή θα πει, μα δεν γίνεται αυτό, έχουμε δικαίωμα να συμμετάσχουμε. Θίξατε ένα καυτό θέμα για τον προπολογισμό, για τα κονδύλια. Θέλω να το αφήσουμε εκτό, διότι αύριο στη συνεδρίαση θα συζητήσουμε σε βάθο το θέμα. Με τα 76% δεν, επαρκώ, δεν επαρκούμε και δεν συμφωνώ. Δεν πάω τόσο μακριά όπως κάποτε παλιότερα. Είμαι πρόθυμη και από τα 90% να μειώσω αυτό το επίπεδο προ όφελο τέλο πάντων των πολιτών. Αλλά θα έλεγα κάπου πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή στο 83-84% να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Αλλά ήδη τώρα σας το λέω, μετά θα ακολουθήσει πάλι γιατί κάποιος το ανέφερε και αυτό, θα έχουμε μια δυνατότητα στο πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί, cross-border διασυνοριακή, πώς το λέμε αυτό, cross-sectoral, διατομεακή συνεργασία που θα μπορεί να διασφαλιστεί και σε ποσοστό να, να καθοριστεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Αύριο. Αύριο θα μπορείτε να το δείτε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Προσεγγίζουμε οι μεν τους δε. Θέλω αυτό που έκανε, αυτό που θέλαμε με το άλλο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το καταστήσει εφικτό, να είναι εφικτό διατομεακά. Το θέλαμε στο παρελθόν, δεν ήταν τότε δυνατόν, εξακολουθούμε να το θέλουμε και θέλουμε ενδεικτικά ελάχιστα ποσά να εγγραφούν που δεν μπορούμε να τα υποβαθμίσουμε και να τα χαμηλώσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να το δεχθούμε αυτό γιατί διαφορετικά δίνουμε μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στους υπαλλήλους της Επιτροπής και δεν γίνεται αυτό. Εμείς είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών. Μας έχουν εκλέξει οι πολίτες λογοδοτούμεναν των πολιτών μας και πρέπει να υπάρξει κατανόηση γι' αυτό και εμείς θέλουμε να καθαρίσουμε αυτό. Η κυρία Νενταλόβα αναφέρθηκε για το πρόγραμμα ε, και για το, την λήξη. Θα ε, πρέπει να ε, δούμε το πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Ο κύριος Μπόρις μίλησε για τον προϋπολογισμό. Έδωσα απάντηση γι' αυτό, τη δική μου μου απάντηση βέβαια. Και το θέμα για την κυρία Μπεναρά Μπατού, για το βουαζινάζ στην γειτονία δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ το πλαίσιο το ευρωμεσογειακό, διότι οι ευρωμεσογειακές χώρες, όπως και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, βρίσκονται στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Έχουμε μια πολιτική γειτονία για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και για τις χώρες του Μεσογείου. Για τη γειτονία αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά και στρέφουμε και προσοχή, με το βλέμμα μας με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και για τις επιθυμίες που θέλουμε να υλοποιηθούν. Έρχομαι στον τίτλο τώρα. Εντάξει. Ευρώπη, Europe, γαλλικά σε αυτό, Europe. Yes Europe, ναι στην Ευρώπη. Αν πούμε Yes Europe παρά είναι γαλλικό. Europe είναι γαλλικό, δεν είναι ε, γερμανικό. Θα λέγαμε Europa. Εντάξει. Μα πώς μπορεί να υπάρξει τέτοια διαφοροποίηση. Πηγαίνετε στους δρόμους του Παρισιού ή οπουδήποτε όλος ο κόσμος ξέρει το yes. Ναι, αλλά όχι ως πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ναι, αλλά θα γίνει ένα πραγματικό όνομα, μάρκα. Ένα γνωστό όνομα, διότι Yes Europe σημαίνει ότι όλοι θέλουμε να βελτιωθεί αυτή η Ευρώπη του Αντενάουρ, του Σούμαν, του Μονέ, του Γκάσπερη, όλων των ίδρυτων Πιστεύω το ΓΕΣ yes είναι πολύ οικείο. Όλοι γνωρίζουν το ΓΕΣ, yes, ακόμη και στη Γαλλία. Εσείς πώς θα το μεταφράζετε το lifelong learning ε, formation, λέει του το Λαβή στα γαλλικά. Ναι, δεν είναι το lifelong learning αυτό, δεν είναι η διαβίου μάθηση. Το μεταφράσατε και θέλετε να το μεταφράσετε και να πείτε we Europe ε, και το yes πώς θα το μεταφράσουμε. Να σας βοηθήσω. Θα σας βοηθήσω εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, σταματάω τώρα και δίνω το λόγο στον κύριο Κορέλ. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα και τους συναδέλφους μου ήταν μεγάλη χαρά να ηγούμε των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα. Ανταποκρίνουμε στην ενδιαφέρουσα πρόκληση και όπως έχω ήδη πει, πιστεύω βαθιά στις προτάσεις βελτίωσης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αυτά που μας ενώνουν. Τα προγράμματα που τρέχουν είναι εξαιρετικά, το θέμα είναι να τα βελτιώσουμε περαιτέρω. Και αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε. Απαντώ σε ορισμένα ερωτήματα. Όσον αφορά τους διδακτορικούς φοιτητές. Τι θα γίνει με τους υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Δύο παραμέτρους πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σήμερα, στο σημερινό έρασμος, το έρασμος όχι το έρασμος μόντους, έχουμε δύο δράσεις οι οποίες θα συνεχιστούν. Κινητικότητα πιστώσεων για τους υποψηφίους διδάκτορες. Χρηματοδοτούμε 3.000 που εποφελούνται από το πρόγραμμα για την κινητικότητα. Αυτό θα συνεχιστεί. Και αν αποδεχτείτε την πρότασή μας, θα είναι ανοιχτό και στην διεθνή κινητικότητα, με τρίτες χώρες δηλαδή. Δεύτερον, όταν λέμε συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, φυσικά ακόμη και σήμερα υπάρχουν προγράμματα τα οποία καλύπτουν και υποψηφίους διδάκτορες και αυτά θα συνεχιστούν στο μέλλον εάν φυσικά γίνει αποδεκτή η πρότασή μας. Θα περιληφθούν στο νέο πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά τα κοινά προγράμματα στο Erasmus Mundus των διδακτορικών, γιατί έχουμε τα κοινά μάστερ και τα κοινά διδακτορικά. Αυτά πέτυχαν όμως ο προπολογισμό δεν ε, είναι ικανοποιητικό. Σήμερα χρηματοδοτούμε περίπου 10 κοινά διδακτορικά. Μόνο. Αυτά σήμερα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το Marie Curie και μάλιστα κάποια τέτοια κοινά προγράμματα όντως χρηματοδοτούνται και ο κύριος Λόκερκαρτ ξέρει ότι το Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Διδακτορικό και αυτό χρηματοδοτείται. Οπότε να διευκρινίσουμε ότι άλλο το μάστερ, άλλο τα διδακτορικά. Δεν μιλώ, προσέξτε, για την κινητικότητα, τα διδακτορικά θα μπορούσαν να πάνε στο Marie Curie. Εκεί θα βρουν χρηματοδότηση και έτσι η εκπαίδευση και η αγορά θα είναι πιο κοντά στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020. Αυτό άλλωστε το θέλουμε να κάνουμε, οι ερευνητές να έρθουν πιο κοντά στην αγορά. Αυτά για τους διδακτορικούς φοιτητές. Το άλλο θέμα το οποίο προέκυψε σαφώ είναι το θέμα των εγγυημένων δανείων. Και προκειμένου να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, μιλούμε για συμπληρωματικό μηχανισμό. Συμπληρώνουμε δηλαδή άλλε υποτροφίε ή το Εράσμος μούντου ή το απλό έρασμο. Αυτά συμπληρώνονται. Απλώς προσθέτουμε μια επιπλέον ευκαιρία στους φοιτητέ, οι οποίοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα μάστερ σε χώρα εκτός της δική του ή εκτό αυτή στην οποία πήραν το πρώτο πτυχίο. Τι εννοούμε όμω όταν λέμε εγγύηση. Δεν εγγυόμεθα το 100% του κονδυλίου που θα καταμιεύσουν οι τράπεζες υπέρ του μηχανισμού. Όχι. Αλλιώ θα ήταν πολύ εύκολο. Εγγυόμεθα 80% το οποίο σημαίνει ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν μερίδιο του κινδύνου, όμως μετριάζουμε τον κίνδυνο κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Πρέπει να λάβουμε συναφώς υπόψη μας την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε μια φορολογική ένωση. Δεν είμαστε μια ένωση τραπεζών. Συνεπώς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια χώρα, ένα κοινωνικό σύστημα αποπληρωμή δηλαδή συναρτήσει των εσόδων του νεαρού επαγγελματία κλπ. Εδώ δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει τέτοιου είδου συντονισμό. Προτείνουμε λοιπόν από τη μία πλευρά ένα καταποκοπήν ποσό αποπληρωμή και κάποιες εγγύησεις για τους δανειζομένους. Προτείνουμε δηλαδή συγκεκριμένα μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια. Προβλέπουμε περίοδο χάριτος, δηλαδή ο δανειζόμενο δεν θα χρειαστεί να αρχίσει να αποπληρώνει παρά μετά την παρέλευση 12 μηνών μετά το τέλος των σπουδών και επίσης λαμβάνουμε υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση του δανειζομένου στην περίπτωση για παράδειγμα οικονομικών δυσκολιών, απώλεια θέση εργασίας, ασθένειας, μητρότητας. Ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει αναστολή της υποχρέωση καταβολής αποπληρωμής του δανείου και βέβαια υπάρχει η ασφάλιση στην περίπτωση θανάτου ή αναπηρία. Επίσης, δεν προβλέπονται, πολύ σημαντικό αυτό, κυρώσει προ αυξήσει, δηλαδή στην περίπτωση πρόορη αποπληρωμής. Αυτό σημαίνει εγγύηση προκειμένου. Πρόκειται λοιπόν για κοινωνικά κριτήρια και κοινωνικά μελήματα. Και βεβαίω το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του φοιτητή και της οικογένειάς του. Η τράπεζα λοιπόν, το μόνο το οποίο θα ζητά από τον φοιτητή είναι απόδειξη ότι είναι γεγραμμένο στην σχετική σχολή για μάστερ. Άρα λοιπόν δεν θα κρίνονται οι φοιτητέ με βάση την οικονομική τους κατάσταση ή το εισόδημα της οικογένειας. Επίσης, δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αντικειμένων των θεμάτων μελέτης, των σχολών. Όλα κρίνονται επίση όρει. Τέλος, η εθελοντική έννοια του μηχανισμού. Εδώ έχουμε ένα μάλλον φιλοσοφικό πρόβλημα, ένα ζήτημα αρχής. Όντως, δεν θα αποφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα αποφεληθούν όλα τα πανεπιστήμια όλες οι χώρες με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι, όπως και να το κάνουμε, θα υποφεληθούν περισσότερο. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για το πρόγραμμα. Για την κατανομή τώρα του προπολογισμού. Ήδη αποδεχθήκαμε το, την πραγματικότητα, του γεγονό ότι οι πολιτικοί θα λάβουν κάποιες αποφάσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση αυτού του προπολογισμού στον γενικότερο προπολογισμό. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία μεταξύ της πολιτικής απόφασης με επαρκή ευελιξία για να ληφθεί η υπόψη, όπως και εσείς το είπατε, τις απρόλεπτες εξελίξεις και την ανάγκη να χρηματοδοτήσουμε διατομιακά προγράμματα. Εννοείται ότι όταν συζητήσουμε την κατανομή αυτών των πόρων κατά τομέα, προσθέτουμε ένα πρόγραμμα, διότι πέρα από το ερασμό, έχουμε το εράσμο μούντού. Άρα η γραμμή του προπολισμού πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε ήταν το ζήτημα των εξόχων απομακρυσμένων εδαφών. Ο, ο ορισμός ε, τώρα του ποια εδάφη καλύπτονται από αυτό τον ε, ορισμό είναι μια απόφαση που έχει ήδη οθετηθεί από το Συμβούλιο Καπολού. Αυτό που βλέπουμε σήμερα με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι το πρόγραμμα ε, εφαρμόζεται σε αυτά τα υπερπόντια εδάφη. Και θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μια τεχνική λύση γι' αυτό αργότερα. Όσον αφορά τον ορισμό των φοιτητών, τι καλύψατε καλύτερα, κυρία Πάκ, από ότι εγώ. Μιλάμε φυσικά για ανθρώπους σε φάση μάθησης ε, παιδείας. Ε, το άρθρο 7 της πρώτης κομισιόν καλύπτει τα όσα καλύπτει ο Λεωνάρδο ήδη. Δεν θα είναι πρόβλημα. Λοιπόν, ένα άλλο σημαντικό σημείο ήταν η επέκταση τη διεθνού συνεργασία στην ε, επαγγελματική κατάρτιση. Παρά τη σπουδαιότητα τη επαγγελματική κατάρτιση για τι αναπτυσσόμενε χώρε, είναι σαφέ ότι με τα χρήματα, με το ποσά που θα εκχωρηθούν στη διεθνή διάσταση του νέου προγράμματο από τους μηχανισμούς εξωτερική δράση καλύπτεται μόνο η ανώτατη εκπαίδευση σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν για να προσθέσουμε την επαγγελματική κατάρτιση να κινητοποιήσουμε κεφάλαια από την κεφαλίδα 1. Τα τελευταία μου δύο σημεία αφορούν την ελεύθερη αγορά ε, και το ζήτημα των 12-15 μηνών θα το κοιτάξουμε αυτό τώρα οι 15 μήνες μπορεί να ε, δημιουργήσουν κάποια τεχνικά προβλήματα διαχείριση του προβλήματος αλλά θα επανέλθουμε σε εσά για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελίξη εδώ όσον αφορά το ζήτημα του αθλητισμού θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι οποιαδήποτε δράση που χρηματοδοτείται από το νέο πρόγραμμα πρέπει να έχει ένα διεθνικό στοιχείο. Διαφορετικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εθνικά κονδύλια. Δεν θα έχει προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ιδρύματα Ζαν Μονέ, φυσικά η συζήτηση είναι δύσκολη. Γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε μόνο δύο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη διότι αλλιώ θα ανοίξουμε το κουτί τη Πανδώρα και θα έχουμε πάρα πολλά ιδρύματα σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την πρόθεσή μας, δεν θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι καλύψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Αν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο, παρακαλώ μην διστάσετε να με ρωτήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημείωσα ότι είπατε, κύριε Κορέλ, ότι πρέπει να σκεφτούμε το Erasmus Mundus τώρα να ενταχθεί στο Erasmus, στο Erasmus. Αληθεύει αυτό. Αλλά ξεχάσατε να πείτε ότι η υποδιδακτορική διατριβή πάνε στο Marie Curie εν μέρη ή όχι. Πού εντάσσονται. Γι' αυτό θα πάνετε εσείς λιγότερα έτσι. Ε, τουλάχιστον να μείνουμε στο πλαίσιο της αλήθειας, να μην λέμε κάποια πράγματα τα οποία δεν αληθεύουν. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό, πείτε μας, ευχαριστώ. Thank you. Ε, ε, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα έχουμε πολύ λιγότερα δοκτορά από ότι μάστερ. Έχουμε 10 διδακτορικά ετησίω από το Erasmus Mundus 2 και έχουμε 35 ετησίω μάστερ από το 2000. Είναι τεράστια διαφορά όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι φυσικά ένα μέρος της χρηματοδότησης ε, των υπαρχόντων κοινών προγραμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται από το νέο πρόγραμμα Γνωρίζετε ότι τα προγράμματα διαρκούν πέντε χρόνια και η χρηματοδότηση θα πρέπει να συνεχίσει υπό το νέο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι του προπολογισμού του νέου προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει προϋπάρχουσες δεσμεύσεις ε, υπό το υπάρχον Ερασμός Μόντους. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα το κομμάτι της χρηματοδότησης που θα μεταβιβαστεί στο Μαρικιουρί θα είναι πολύ μικρό, αλλά με τη μεταβίβασή του στο Μαρικιουρί θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο Μαρικιουρί και έτσι θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε πολύ περισσότερα διδακτορικά. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορέρ. Να επιστήσω την προσοχή στο εξή. Αν προσέξατε και ακούσατε προσεκτικά, ο κύριος Κορέλ με σαφήνεια αναφέρθηκε και εξήγησε το θέμα των loan facilities και πολλά από αυτά που περιέχονται στις τροπολογίες έχουν συμπεριληφθεί στις παρατηρήσεις και τα, στα όσα είπε. Και ελπίζω Τουλάχιστον θα κάνω την δική μου συμβιβαστική πρόταση όταν θα έρθει η ώρα να την κάνω. Αυτά τα οποία προανέφερε ω προπόθεση θα τα χρησιμοποιήσω. ω όρο και προπόθεση. Την δομή που μα περιέγραψε θα την ε, συμπεριλάβω στη συμβαστική μου τροπολογία. Αυτή η δομή θα πρέπει να γίνει νόμο. Στο κείμενο θα αναφέρεται ω νόμο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριο Λόκεγκαρτ, παρακαλώ, μια ερώτηση είχε. Ναι, απλά μια, ένα μικρό σχόλιο για αυτές τις εγγύησεις δανείων. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι κατάλαβα τα σχόλια και του κύριο Κορέλ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι σωστά. Αυτό που με ανησυχεί μόνο είναι ότι κάποια στιγμή εμείς ξεκινήσαμε διαπραγματεύσαμε το Συμβούλιο ως Σοφό θα ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει να εισάγουμε αυτό το σύστημα εγγυήσεων δανείων να λάβουμε υπόψη ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θα κέρδιζαν τίποτα από αυτό. Είναι λοιπόν ένα πολιτικό ζήτημα αυτό. Αν θέλουμε την υποστήριξη ευρεία συνένεση εντός του Συμβουλίου και παραδέχομαι είναι πολύ ιδεαλιστικό αυτό το σύστημα εγγύησης δανείων. Το υποστηρίζω προσωπικά, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς γι' αυτό. Είναι και ένα πολιτικό ζήτημα και ορισμένα κράτη-μέλη σαφώς υποστηρίζουν το πρόγραμμα Εράσμους αλλά έχουν κάποιους συνδυασμού για αυτό το ζήτημα Σα Καλό λοιπόν να το λάβετε υπόψη αυτούς τους συνδυασμού. Ναι, το κατανοώ πολύ καλά αυτό που είπατε, αλλά και πιο πριν το είπα. Αν τώρα σκεφτούμε άλλες χώρες, που δεν έχουν φοιτητέ στο πρόγραμμα έρασμο. Ε, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει, υπήρχε. Αν κάποιο δεν μπορεί να συμμετάσχει, δεν μπορεί να υποχρεωθεί και θέλουμε με αυτή την προσφορά, δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε κανέναν. Το πρόβλημα όμω είναι ότι η Δανία, για παράδειγμα, είχα πάει στο Όρχιου και με του καθηγητέ από κοινού συζήτησα για αυτό το θέμα. Ότι φυσικά οι Δανείοι μπορεί να πούν «Ε, δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα το κάνουμε εμεί οι ίδιοι». Το λένε και οι Γερμανοί αυτό αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον πρέπει να έχουμε αρκετή αλληλεγγύη που θα εκφράζουμε ώστε για τρεις ή τέσσερις που ίσως δεν θέλουν να το κάνουν να μην ε, θεωρείται ότι είναι κατά του προγράμματος και σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Εκπρόσωποι του Συμβουλίου, παρακαλώ σας παρακαλώ να μας πείτε για αυτό το θέμα δύο λόγια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τον λόγο. Η Κυπριακή Προεδρία θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις συζητήσεις που γίνονται στο Κοινοβούλιο σχετικά με το νέο πρόγραμμα και όπως επανελειμμένα έχουμε τονίσει σημασία ουσιαστικά ε, είμαστε ανοιχτοί σε μια ειλικρινή συνεργασία για να οδηγήσουμε τις διαπραγματεύσεις σε μια ευτυχή κατάληξη προς το συμφέρον των νέων και όχι μόνο των νέων της Ευρώπης und lassen Sie mich ε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τώρα τη γλώσσα της Προέδρου. Η Επιτροπή Πολιτισμού του Συμβουλίου σε μία από τις συνεδριάσεις της το σχέδιο της έκθεσής σας το έλαβε υπόψη και αναμένει τώρα την ψήφιση στις 26-27 Νοεμβρίου που θα ψηφιστεί που με το Συμβούλιο Υπουργών Συμπίπτη, Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας και Αθλητισμού. Όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο έχει ε, μια κοινή κατεύθυνση σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθόρισε με κοινή κατεύθυνση. Μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι σε πολλά σημεία υπάρχει συμφωνία όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο για, τους, για την νεολαία, για τους νέους, για τη διατήρηση των έξι αυτών ε, ιδρυμάτων μέσω του Ζαν Μονέ για την ελαστικότητα όσον αφορά τις εθνικές υπηρεσίες και οργανώσεις και σε συμφωνία με τις εθνικές πρακτικές φυσικά και σε κάποια άλλα σημεία επιπλέον επίσης. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι τομείς όπου εμείς λιγότερο συμφωνούμε. Εντάξει, με κάποιες προτάσεις, όπως για παράδειγμα με το μεγάλο αριθμό των νέων επιπρόσθετων στόχων που το κείμενο σε κάποια σημεία, πώς να το πω, το καθιστούν ασαφές ή θα μπορούσαν να το καταστήσουν ασαφέστερο σε σχέση με τα πλαίσια αυτά. Όπως γνωρίζετε πρόεδρε, εμπεριέχονται σε αυτές τις κοινέ κατευθύνσεις του Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται όλα και άπαντα τα σημεία που με τον ένα ή άλλο τρόπο εξαρτώνται από κονδύλια του προϋπολογισμού. Ένα από αυτά, όπως εσείς είπατε και ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το νέο προτινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω για την χρηματοδότηση, μέσω διευκόλυνσης δανείων πιστώσεων για φοιτητές μάστερ. Η Προεδρία αυτό το θέμα δύο φορές το ενέγραψε στην ημερήσια διάταξη των Υπουργών Παιδείας ακόμα και σε άλλες συνεδριάσεις ε, πρόκειται να συζητηθεί εκ νέου. Στόχος μας είναι με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσουμε σαφήνεια για αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο. Ούτε απορρίπτουμε ούτε υποστηρίζουμε, μια και δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πώς θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Και ποιες επιπτώσεις θα έχει ή θα μπορούσε να είχε κάτι τέτοιο. Και περαιτέρω θα προσπαθήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες και εναλλακτικέ δυνατότητες λειτουργίας του νέου μέσου να τις ε, εντάξουμε ή να μπορέσουμε να τις εντάξουμε και να τις κατοχυρώσουμε σε ένα σαφές πλαίσιο. Για την περίπτωση, το τονίζω, για την περίπτωση που το μέσο αυτό εγκριθεί τελικά. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Πρόεδρε, και χαιρόμαστε για την επικοδομητική γόνιμη συνεργασία. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Συμβούλιο είδατε το ότι εμείς ε, το έργο που κάνατε το ακολουθήσαμε και σε κάποια σημεία βρέθηκε συνένεση με σας. Και τώρα η Ευρω... εμείς, εμείς, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα με τη νέα πρόταση που θα υποβάλουμε, τον συμβιβασμό που θα υποβάλουμε για το loan facility, θα σας δώσουμε ευκαιρία να πείτε ναι και να εγκρίνετε συμβούλιο θα έλεγα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται που και εσείς ε, αναφέρατε και ζητήσατε και θα θέλατε και εμείς το ίδιο εργάστηκε και επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα μια και είχαμε τόσες πολλές τροπολογίες και αυτό ήταν και προς το δικό σας νομίζω ε, συμφέρον Παρακαλώ να μην πιστέψετε ότι κάτι θα κάνουμε ασαφέστερο. Το αντίθετο δεν θα γίνει κάτι ασαφέστερο αλλά σαφέστερο. Έχουμε προσδιορίσει κάποιους στόχους και τους έχουμε αποσαφηνίσει. Το χαρτί είναι υπομονετικό όμως. Είναι πολύ ε, υπομονετικό και δεν εμποδίζει κανέναν να κατανοήσει τα πράγματα. Το αντίθετο κιόλα. Κάθε ένας που έχει συμφέρον και ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα να δει τι θα γίνει με αυτά τα προγράμματα, τι θα υποστηριχθεί. Αν έχουμε μόνο γενική συνεργασία ως τίτλο, είναι πολύ λίγο αυτό, πενιχρότατο. Πρέπει κάτι παραπάνω να αναφέρεται. Στο αίτημα των φιλελευθέρων από πλευράς του συναδέφου Λόκεγκαρτ, ακολουθώντας το αίτημα αυτό, το κάναμε, συμπτύξαμε περισσότερο για να είναι πιο αποτελεσματικό. Υποβλήθηκε και μια συμβαστική πρόταση ως τροπολογία. Μπορούμε να συνενέσουμε, να προσεγγίσουμε ένα τον άλλο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και εσείς να πιστεύετε ότι στους πολίτες ή σε εκείνους που έξι χρόνια θα μπορούν ή θα πρέπει να εργαστούν με αυτά, θα πρέπει να τους πούμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο υπήρξε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο ή μακρύτερο πλαίσιο. Αλλά εδώ υπήρξε σύνμηση μετά την παρέμβαση της Επιτροπής, τη θέση της Επιτροπής, προσεγγίζουμε ένα τον άλλο. Είναι πολύ καλό να συνεργαζόμαστε μαζί. Αν σκεφτούμε πώς ξεκινήσαμε, με χαρά μπορώ να πω ότι προσεγγίσαμε πολύ ο ένας τον άλλον. Και έτσι λοιπόν δεν πρέπει να ε, φοβόμαστε. Μέχρι τον τριμερή διάλογο ευελπιστώ ότι και άλλα εμπόδια θα έχουν αρθεί. Διότι ένα είναι κοινό για όλους μας είναι συμφέρον μας η επόμενη γενεά να εκπαιδευτεί και να καταρτιστεί καλά, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα στα χέρια μας στην Ευρώπη. Οι καλά εκπαιδευμένοι νέοι είναι το μέσο, το εργαλείο μας. Εκεί πρέπει να εργαστούμε. Το Συμβούλιο καλό θα ήταν με, τη μεσοπρόθεσμη, με το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό ή προγραμματισμό για τα κονδύλια που θα διαθέσει να σκεφτεί να μην περικόψει κονδύλια. Τα λίγα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μπορεί οι περικοπές να γίνουν αλλού και όχι από αυτά τα κονδύλια που μας διαθέτεται. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι πολλά αυτά τα λεφτά. Στα μεγάλα προγράμματα δεν θα τα κατονομάσω ποια είναι για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Αν όμως πάρετε από παντού κάποια κονδύλια και τα δώσετε σε αυτό το πρόγραμμα, τότε αυτά τα οποία προβλέφθηκαν από την Ευρωπαϊκή θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Χρειαζόμαστε αυτή την αύξηση για τη στρατηγική του 2020 για να πλησιάσουμε τους στόχους μας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να παρεκκλίνει και να σκέφτεται κάτι διαφορετικό. Ίσως οι Υπουργοί Οικονομικών. Αλλά δεν επιτρέπεται εκείνοι να αποφασίζουν όλα και τα πάντα ε, λοιπόν, τότε όταν λένε ότι δεν υπάρχουν περισσότερα χρήματα, εκείνοι που θέλουν να εργαστούν περισσότερο, να εργαστούν για τα παιδιά. Να ξέρουν ότι αν εξοικονομήσουν σε αυτά τα προγράμματα, δεν πρέπει να εξοικονομήσουν στα δικά μα προγράμματα για την εκπαίδευση και παιδεία και κατάρτιση. Όχι επειδή είμαστε ωραίοι και καλοί, αλλά επειδή είναι απόλυτα αναγκαίο για την παιδεία και εκπαίδευση να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει περισσότερο. Θα είχαμε λιγότερη ανεργία στην Ισπανία, αν π.χ. στην Ισπανία γινόντουσαν περισσότερα για την εκμάθηση γλωσσών από τους νέους. Αν είχαν μάθει γερμανικά περισσότεροι νέοι στην Ισπανία θα μπορούσαν να εργαζόντουσαν περισσότεροι από αυτούς στη Γερμανία που υπάρχουν θέσεις για να απασχοληθούν. Αλλά δεν έγιναν αυτά. Να μην περικόψουμε λοιπόν αλλά να αυξήσουμε τα κονδύλια και έτσι από κοινού θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα κατανείμουμε αυτά τα ποσοστά χωρίς ε, να αφαιρεθούν εξουσίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ο κοινό στόχος μας θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Και έτσι ολοκληρώνω αυτή τη συζήτηση. Εδώ ολοκληρώνεται. Ευχαριστώ ρητά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και τους συναδέλφους για μια καρποφόρα γόνιμη καλή συνεργασία. Και αύριο νωρί μέχρι το μεσημέρι θα έχετε τις συμβαστικές μου τροπολογίες για το προϋπολογισμό, για το, τα αθλήματα και για τη διευκόλυνση για τα δάνεια. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης τώρα. Περνάμε στο σημείο 7 και στο σημείο 8, μια και είναι και από τον ίδιο εισήγητη που έχουν εκπονηθεί. Και επειδή υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους, Πρόκειται λοιπόν για την ευθύνη, για την προαγωγή των ε, ε, δράσεων των συμφερόντων της κοινωνίας, για την προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας στην πορεία προ βιώσιμη ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς και ο τίτλος ε, για τη δεύτερη δεν θα τον επαναλάβω. Τον Οκτώβριο του 2011 είχε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεωμένη στρατηγική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινωνική εταιρική ευθέρη, ο κύριο, ε, ευθύνη. Ο κύριος Λόκεγκαντ είναι εισηγητής μας. Συνέταξε μια γνωμοδότηση για αυτό το χαρτοφυλάκιο, για αυτό το θέμα. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Νομικών και Απασχόλησης, Γιούρι και Εμπλ έχουν μη νομοθετικές εκθέσεις που έχουν εκπονήσει για αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έκαναν αυτό υπό το άρθρο 50, Rule 50, περιβόητο άρθρο 50, όπου οι δύο συνεμπλεκόμενες συναρμόδιες επιτροπές μπορούν έτσι να συνεργάζονται. Και έτσι λοιπόν έχουμε εδώ μια γνωμοδότηση από πλευράς μας που μετά μετά την 18 η Δεκεμβρίου για αυτές τις, από αυτές τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές, σε αυτές τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές αποστέλλεται. Ο κύριος Λόκεγκάντ έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ ξανά Πρόεδρε. Ευτυχώς ε, δεν χρειάστηκε να συντάξω δύο γνωμοδοτήσεις αλλά μόνο μία θα είμαι σύντομος καθώς όλοι έχετε τα έγγραφα μαζί σας. Έχω εστιαστεί σε τρία στοιχεία στην γνωμοδότησή μου. Την προβολή, τις ε, πτυχές της παιδείας φυσικά, αφού είμαστε η Επιτροπή Αρμόδια για αυτό και η δυνατότητα χρήσης της έτε ε, στις επιχειρήσεις ε, όταν εργάζονται σε αυτές φοιτητές ως μαθητευόμενοι. τώρα, όσον αφορά τι αναπηρίες και την ευαισθητοποίηση, το στοιχείο νούμερο ένα είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία και οι πολίτε να είναι ευαισθητοποιημένοι για την ΕΤ και το ρόλο που παίζει σε σχέση με την κοινωνία. Εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλλουμε, να κοινοποιούμε, να δημοσιοποιούμε την ΕΤΕ. Όσον αφορά τις πτυχές ε, της εκπαίδευσης, πιστεύω είναι σημαντικό η εταιρική κοινωνική, ευθύνη να συμπεριλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε τόσο οι φοιτητέ όσο και οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ε, ότι δυνατό περισσότερο σε σχέση με την ΕΤΕ ε, μετά. Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουν οι φοιτητέ εμπειρία για αυτό το θέμα κατά τις σπουδέ τους. Είναι ένα εργαλείο που μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ε, κατά τις περιόδους μαθητείας. Και ελπίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται καλά στη γνωμοδότησή μου. Αναμένω τα σχόλιά σας. Και φυσικά αν υπάρξουν προβλήματα μπορούμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση παρότι δεν, περιμένω, δεν προβλέπω να γίνει κάτι τέτοιο γιατί το ζήτημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αντικρόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σιλβία Κώστα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ για αυτά τα σημεία που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Λάκεγκαρτ. Ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Θα δώσουμε φυσικά και τροπολόγιες. Ε, όσον αφορά τις σχέσεις επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, έχουμε εμπειρίες καλών σχέσεων και στην Ευρώπη και στη χώρα μου μεταξύ των ε, τελευταίων ετών των πανεπιστημίων και των λυκείων και δυνατότητες ε, μερικών ωρών εμπειρίας ε, επαγγελματικής κατάρτισης. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο αλλά και τα τελευταία έτη του Λυκείου. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό που υπογραμμίσατε την απέτηση οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν περισσότερο τον αθελοντισμό, την πραγματική δυνατότητα ε, εθελοντικής εργασίας στις επιχειρήσεις και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί και αντικείμενο εθνικών συμβάσεων εργασίας να αναγνωρίζεται όπως ορισμένα κράτη-μέλη η δυνατότητα μορφός, μορφών απουσίες για θελοντική εργασία, το οποίο αναγνώριζεται και ως δικαίωμα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, αλλά και αναγνώριση επίσημων και άτυπων προφίλ αρμοδιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον, γνωρίζω εμπειρίες πολύ ενδιαφέρουσε, για άτομα που έκαναν εθελοντική εργασία σε ορισμένε, πεφωτισμένε τράπεζε που υιοθέτησαν ένα τέτοιο σύστημα και αναγνώριζαν το έργο που επιτέλεσαν οι εθελοντές εκεί. Το άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω ως ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα προώθησης και μέσω των δικτύων του Aerobusiness, τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια κτλ. Δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να εντοπιστούν οι βέλτιστε πρακτικέ ε, και να ενισχυθεί η πεποίθηση ότι εδώ πρόκειται για μια νέα διάσταση με τον οποίο μια, επιτελεί μια επιχείρηση το ρόλο της, δηλαδή όχι μόνο profit for profit, όχι μόνο δηλαδή για το κέρδος, αλλά και ένα κοινωνικό ρόλο. Ευχαριστώ. Vielen Ευχαριστούμε πολύ. Τα σχόλια που μόλις προσέθεσε η κυρία Κώστα υπάρχουν ήδη μέσα στο κείμενο. Το, στο σημείο 4 αναφέρονται τα σχολεία και οι μαθητές σχολείων και οι επισκέψεις σχολείων υπάρχουν στο σημείο 4. Μάλιστα, ήρθε ένας μαθητής σχολείου στο δικό μου γραφείο και μου ζητήθηκε ένας 16χρονος μαθητής να έρθει να επισκεφτεί το γραφείο μου και ήταν καταπληκτικό το να βλέπει κανεί ε, πόσο απορρόφησε ο, τα πάντα αυτός ο μαθητής ε, ό,τι συνέβαινε εδώ πέρα και όπως φαίνεται στη χώρα μου υπάρχουν πολλές συνεργασίες μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων ε, στη Γερμανία και μάλιστα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς ε, είναι ήδη κάτι που γίνεται αλλά και που θα πρέπει να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο. οικονομική δέσμευση τώρα ε, περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 6, η ανάπτυξη και όλα αυτά στο κεφάλαιο 6. Θα μπορούσαμε ίσως να το καταστήσουμε λίγο πιο σαφές, να το παρουσιάσουμε πιο καθαρά. Ε, θα μπορούσατε να επιβάλλετε μια τροπολογία γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι όσα είπατε περιλαμβάνονται εδώ, αντικατοπτρίζει τα όσα είπαμε στην αρχή. Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Το τονίζουμε διαρκώς πόσο απαραίτητο είναι αυτό. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε με τα όσα είπατε θα μπορούσαν ίσως να διατυπωθούν με λίγο μεγαλύτερη σαφήνεια, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο για τροπολογίες μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, τις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Μόρτεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το θέμα ή πιστεύεις ότι υπόθηκαν όλα. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι υπόθηκαν όλα. Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε ε, λοιπόν, τα σημεία 7 και 8 ολοκληρώθηκαν. Έτσι φτάνουμε στο σημείο 9 τη σημερινή διάταξη εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωση για την νεολαία 2010-2012. Δίνω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου. Παρακαλώ. Thank you, Madam ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή για την ανακοινωσή τη. Θα είμαι σύντομο, αλλά ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω μια γενική, ένα γενικό σχόλιο ότι καθώς θεωρούμε δεδομένο ότι η στρατηγική, η κοινή στρατηγική για την νεολαία είναι κοινή, ενιαία και ότι δεν ε, χωρίζεται σε πολλές διαφορετικές πρωτοβουλίες, Φυσικά καθώς αυτή η Επιτροπή είναι κατά κάποιο τρόπο η πρωτεύουσα, η, σημαντική, η επί Επιτροπή, χρειαζόμαστε μια διατομαϊκή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την νεολαία. Γι' αυτό θα αναφέρω τρία στόχευμένα ζητήματα ως γενική εισαγωγή σήμερα, χωρίς να αναφερθώ σε λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν αναφέρει το Συμβούλιο, Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι που η Κομισιόν στην ανακοίνωσή τη ακολουθεί την ίδια προσέγγιση. Έχοντα αυτά υπόψη, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ ειλικρινή. Πριν, πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία, που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε του νέου. Και θεωρούμε ότι βοηθάει του νέου ανθρώπου θα προσέθετε σε αυτούς προς τη θέμενη αξία το ίδιο και στην ευρωπαϊκή κοινωνία γενικότερα. Φυσικά συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να υποστηρίζουμε περισσότερο και να είμαστε πιο παραγωγικοί. Από τότε όμως, και αυτό πρέπει να το αναφέρω, η κατάσταση άλλαξε, επιδεινώθηκε δραματικά η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης, επηρέασε την νεολαία με απροσδόκητο τρόπο, αυξήθηκε η ανεργία στο 23% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία των νέων σε ορισμένα κράτη-μέλη όπως στην Ελλάδα και την Ισπανία έχουμε φτάσει στο 76-77%, 35% στην Ιταλία και στη Γαλλία ακόμα έχουμε ανεργία νέων σε επίπεδα 26%. Από την άλλη πλευρά, περίπου το 17% των νέων δεν ε, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις νέους σήμερα δεν κάνει τίποτα. Δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ως Ευρώπη, το έχουμε συζητήσει όλο αυτό. Στην ίδια περίοδο από το 2010 μέχρι σήμερα περιόρισαν τις δαπάνες ε, στην εκπαίδευση όλα τα κράτη-μέλη, έως ε, και στο 10% το 2020 στοχεύει σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε επίση ότι η στρατηγική για την νεολαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να υλοποιείται προ το ήμουν δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό που θα προσπαθήσω να τονίσω είναι ότι θα ήθελα αυτή η έκθεση να έχει περισσότερες από μία σελίδες αφιερώμενες στις επιπτώσεις της κρίσης τους νέους στην ανακοίνωση και πιστεύω ότι εάν παραμείνουμε επικεντρωμένοι σε αυτή τη σελίδα αν παραμείνουμε στο κείμενο που έχουμε σήμερα είναι σαν να δείχνουμε σε όλους τους πολίτες μας, σε όλους τους συντελεστές που μας παρακολουθούν ότι είμαστε μακριά ανοιχτομένοι. Δεύτερη παρατήρηση. Στην περίοδο από το 10 έως το 12 έλαβαν χώρα τεράστιες αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των νέων για πολλού. τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν υπεύθυνα για πολλά δεινά. Είχαμε επαναστάσεις ε, στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικών δικτύωσης που αποτέλεσαν για ορισμένους σημαντικό παράγοντα για την Αραβική Άνοιξη. Πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων συμμετέχουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση και δεν αφιερώνουμε σε αυτά καμία παράγραφο σε αυτή την έκθεση. Πριν από τρία χρόνια σε αυτή την Επιτροπή στο σχετικό θέμα ε, για τους νέους επιμείναμε για δείκτες, για αξιολόγηση προόδου, παρακολούθηση στο πλαίσιο και της ανοιχτή μεθόδου συντονισμού και συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού. Αναφερόμαστε στην παράγραφο 4.2 αυτής της έκθεσης, αλλά πιστεύω ότι όσον αφορά τη σύνδεση του κοινή οργάνωση συντονισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Αυτό δεν το ζητάμε χωρίς λόγο το ζητάμε, διότι τα μέλη του Κοινοβουλίου μας συχνά έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα των νέων μας απασχολούν ιδιαίτερα και έτσι έχουμε μια βαθιά γνώση του θέματος που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νέοι της. Και πιστεύουμε ότι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής. Επιμένω σε αυτά τα τρία σημεία, διότι από την ανακοίνωση της Επιτροπής αποκτώ την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε περισσότερα για αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά χρειαζόμαστε περισσότερα. Δεν είναι κρίσιμη αυτή η προσέγγιση της... Ε, δεν επικρίνω αυτή τη στιγμή την Κομισιόν, επικρίνω την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όπως είπα στην αρχή, προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και ε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε φυσικασμένοι με τη σημερινή κατάσταση που αφορά την νεολαία, τα προβλήματα και τις ανάγκες των νέων. Τώρα για να μιλήσω λίγο για το κείμενο της Κομισιόν. Άλλο ένα, ένα πράγμα που ακόμη προσπαθώ να καταλάβω όσον αφορά τι ανακοινώσει τη Κομισιόν για την νεολαία είναι πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει παρέχοντα αποτελέσματα σύμφωνα με τη διατομιακή προσέγγιση στην οποία αναφερόμαστε διαρκώ είναι, δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί σε αυτή την ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στην πρωτοβουλία ευκαιριών για τους νέους που παρουσίασε στις 20 Δεκεμβρίου πέρυσι ο κύριος Μπαρόσο στο πλαίσιο του προγράμματος για τους νέους. Ε, αν δεν απατώμε, τότε μίλησε για ένα δισεκατομμύριο ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η Κομισιόν. Τι έγινε με αυτό. Τότε μίλησε επίσης η Κομισιόν για τη ε, πρώτο γιούρες για μια ιστορία επιτυχίας που ήθελε υποστήριξη υποστηρίζεται επαρκώς ε, βλέπω να γίνεται αναφορά σε αυτή την έκθεση ε, από την Κομισιόν αλλά θα ήθελα περισσότερα όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα επιπλέον σε αυτή την ανακοίνωση δεν αναφέρεται τίποτα για τις ειδικές task force για την νεολαία Είναι άλλη στρατηγική για την νεολαία αυτή. Δεν, δεν έχει μια στρατηγική με συνοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Αυτό προσπαθώ να πω. Θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση από την Κομισιόν. Αυτή η προσέγγιση της Κομισιόν είναι διαφορετική από εκείνη της μονάδας της κυρίας Βασιλείου. Ελπίζω να λάβω μια απάντηση γι' αυτό σήμερα. καθώς έχουν αλλάξει οι περιστάσεις από το 2009 και 2010 πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές. Ε, Γι' αυτό σας έκανα αυτή την παρουσία. Σήμερα θα χρειαστεί να είμαστε πιο ε, να κινητοποιηθούμε περισσότεροι και να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Λυπάμαι που λέω ότι εγώ πιστεύω ότι και όσα συζητήθηκαν το 2010 δεν υλοποιήθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί. Παρατηρώ θετική προσέγγιση στην έκθεση από την Κομισιόν, αλλά πιστεύω ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από το 2010. Ακόμη και οι εμβληματικέ πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τόση επιτυχία παρουσιάζουν προβλήματα. Σα υπενθυμίζω όταν συζητήσαμε πριν δύο εβδομάδε στην Ολομέλεια το πρόγραμμα Εράσμου. Σα υπενθυμίζω επίση τι προσπάθειε τη Επιτροπή μα με την πρόεδρό μας, για, με την πρόεδρό μας ε, για αυτό το νέο ενοποιημένο YES, το πρόγραμμα YES για την διαβίου μάθηση. Αλλά το 2010 Παρακολουθώντας βάσει μελετών την υλοποίηση, πιστεύω τα αποτελέσματα, η υλοποίηση αυτή δεν ήταν επιτυχής. Και αυτό δεν το λέω επειδή δεν πιστεύω στις προσπάθειες ε, της Επιτροπής. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη έχουν τεράστιο, ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη και αυτό που προσπαθώ να πω σήμερα ως εισαγωγή σε αυτή τη νέα έκθεση που προσπαθούμε να έχουμε ως προ, έκθεση πρόοδου της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα. Φυσικά καλωσορίζουμε τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, καλωσορίζουμε επίσης και τη γνωμοδότηση της παρούσα που έχουμε σε αυτή την Επιτροπή από την Επιτροπή Απασχόλησης, είναι κάτι που χρειαζόμαστε, η ανεργία μεταξύ των νέων και τα ποσοστά ενεργείας μεταξύ των νέων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά φυσικά θα χρειαστεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να έχουμε μια ολιστική καθολική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία. σε θέματα απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση όσο και περιβάλλοντο, ε, συμμετοχή ε, στα κοινωνικά και υγεία. Όλοι συμφωνούμε για αυτά τα ζητήματα, αλλά μεταξύ άλλων πρέπει να προτείνουμε και πολιτικέ που θα βοηθούν στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων απασχόληση, ώστε να δράσουμε το ταχύτερο δυνατό και να ανοιχνεύουμε τι περιπτώσεις πρόορη εγκατάλειψης των σχολείων, να παρέχουμε συμβουλές για όσους εγκατέλειψαν τα σχολεία και αναζητούν εργασία. Να υποστηρίξουμε τις δυνατότητες μαθητεία, συνδυασμού μαθητεία και εργασία και μελετών και, να... και μελέτης και ε, σπουδών. Δεν έχω πολλά να πω αλλά δεν θα συνεχίσω διότι γνωρίζω ότι είστε όλοι κουρασμένοι και ενεργά ήδη και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε να το συζητήσουμε στι επόμενε μα ε, συναντήσει, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση όσο έχει ο, αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία στην Ευρώπη δεν μπορούμε να λέμε στην εκθεσή μας ότι δύο χρόνια μετά τη στρατηγική για την νεολαία, δηλαδή δύο χρόνια μετά ε, από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, έχουμε θετικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Εγώ πιστεύω ότι οι εξελίξεις είναι αρνητικές και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Θα χρειαστεί να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί στο τι ζητάμε σε αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι χρειάζεται να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα αυτό και να παρέχουμε κίνητρα για όλα τα κράτη-μέλη, οποιονδήποτε παράγοντα ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ώστε να εφαρμόσουν τα, να δημιουργήσουν τα απαραίτητα σχέδια, διότι η παρούσα γενιά είναι σε κίνδυνο. Και όπως λέμε όλοι, κινδυνεύει και το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ και ξανά. Ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτή την έκθεση και για την ευκαιρία που μας παρέχουν να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και πάλι σε αυτή την Επιτροπή και πιστεύω ότι την παρούσα εποχή με τα μηνύματα που μπορούμε να δώσουμε με μια έκθεση πρωτοβουλίας, ίσως και κάποιες επιπλέον ιδέες, ίσως ένα έτος για την νεολαία, έχουμε κάποιες ιδέες, θα τις συζητήσουμε με τους κοιόδης κάποιες άλλες προσεγγίσεις ε, όπως τη διατομιακή προσέγγιση να χρησιμοποιήσουμε, για να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το 1 δισεκατομμύριο που είναι διαθέσιμο από το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται από Ευρωπαίους ηγέτες και ανώτατα στελέχη ε, πιστεύω ότι έχει να παίξει σημαντικό ρόλο η παρουσία. επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υπομονή σας κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Γιώργο, δεν ήταν πολύ, πώς να το πω, δεν ήταν πολύ ωραίο. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Πιστεύω ότι περιέγραψε στην πραγματικότητα, όπως χρειάζεται καμιά φορά. Δεν πρέπει να έχουμε μόνο ωραία λόγια κατήχησης, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά σωστά. Και για το αν πρέπει ή όχι να κατηγορηθεί η Επιτροπή, ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνο, ο ένοχος. Το Συμβούλιο δεν είναι πλέον εδώ, αλλά είναι το Συμβούλιο υπεύθυνο, ο υπεύθυνο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Νεβενταλόβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν συντομότερη και περιεκτικότερη. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον κύριο Παπα-Νικολάου ήταν θετικό να συνεργαστώ μαζί του γιατί είναι παίων σε σχέση με τα θέματα για την νεολαία και προσπαθούμε για τους νέους να πετύχουμε ό,τι καλύτερο κοινό συμφέρον και στόχος μας. Τώρα θέλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα για την αναγνώριση σε σχέση με τον κέριο ρόλο αυτών των στοιχείων και φυσικά την αναγνώριση των νέων και των οργανώσεων νέων για οποιοδήποτε διάλογος πρέπει να λαμβάνει υπόψη και συμπεριλαμβάνει τις οργανώσεις και συλλόγους νέων. Είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο βήμα αυτό και σε σχέση με την συνεργασία αυτή προσπαθούμε στο Κοινοβούλιο να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις νέων και δίνεται αγώνας ε, για αναβαθμισμένη ποιότητα και φυσικά θέλουμε να έχουμε καλύτερη ζωή για τους νέους μας. Έχουμε διαρθρωμένο διάλογο, είναι καλό να έχουμε συζητήσεις, αλλά πρέπει και το βήμα μετά τις συζητήσεις να ακολουθεί. Αναφέρθηκε μόλις πιο πριν, οι πραγματικές δραστηριότητες και η πραγματικότητα είναι εκείνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μετά τους διαλόγους. Αυτό είναι αυτό που απουσιάζει ακόμα. Δεν έχουμε αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες και λήψη αποφάσεων επαρκώς μετά από τους διαλόγους μετά από τι επαφέ. Επίση, καλό είναι ότι θέλουμε να ενταχθεί το θέμα των νέων στι πολιτικέ youth mainstreaming. Ένα παράδειγμα για συζήτηση για τα προγράμματα για τα επόμενα 7 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θέλουμε να ενταχθούν στα προγράμματα τα θέματα των νέων. Αλλά είναι αργά τώρα να υποβάλλονται τώρα προτάσεις για το youth mainstreaming στα προγράμματα. Καλό είναι αυτό, αλλά στην αρχή πρέπει να γίνεται και να τα σκεφτόμαστε έγκαιρα. Και είναι αυτό κάτι που θα ήθελα να πω από πλευρά μου, το θεωρώ σημαντικό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα τρία χρόνια οι ιδέες που εμπεριέχονται για την κοινωνική ένταξη, κυρίως για την υγεία και την ευεξία των νέων, θετικές ιδέες αυτές και τις καλωσορίζω. Πρέπει να εμπλακούν περισσότερο οι νέοι, να τους εμπλέξουμε. Η κοινωνική ολοκλήρωση, και η κοινωνική ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για το μέλλον και προσωπικά πιστεύω τα θέματα υγείας, η αναπαραγωγική υγεία και τα θέματα επιλογής των νέων μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι νέοι αυτοί και πρέπει να σκεφτόμαστε και να σκεφτούν και το μέλλον τους. Πολύ σημαντικό για τη ζωή τους. Χαίρομαι πολύ αγαπητέ συνάδελφοι να συνεργάζομαι μαζί σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά επαΐων είστε σε αυτά τα θέματα για τους νέους. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κάποια πίκρα που ακούστηκε, μια πικρία και απορρέει φυσικά ίσως από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Κυρίως ενώ την υψηλή ανεργία και την ανικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υψηλής αυτής ανεργίας των νέων. Πώς δηλαδή θα μπορούσαν να απασχοληθούν αυτοί ε, και Πρόκειται για πολύ θετικού νέου ανθρώπου που πρέπει να έχουν ευκαιρίε. Η κρίση όμω είναι αμήλικτη και πλήττει αλήπητα του νέου. Θα έπρεπε ίσω να προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε. Εργαζόμαστε και για τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ μέχρι το 2020. Πρέπει ίσω ένα φόρουμ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων να δημιουργηθεί. Τι θα γίνει στο μέλλον με όλα αυτά τα θέματα και πώ μπορούμε να συντονίσουμε όλα τα προγράμματα και τα μέτρα ώστε η πολιτική για του νέου να έχει καλύτερα πιο θετικά αποτελέσματα για τη στρατηγική ως χρονορίζοντα του 2020 στοχοθετημένες πολιτικές προανήγγειλε πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κ. Μπαρόζο μέτρα για τους νέους, ε, κατάρτιση, εκκινώντας από τη σημερινή πραγματικότητα στην αγορά ε, όπως ισχύουν τα πράγματα σήμερα και το έρασμος ε, όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι μια κίνηση, ένα σημείο κίνηση σε αυτό το σημαντικό πεδίο Πολιτική για τους νέους, ακριβώς με την πολιτική των νέων δημοσιονομικών προοπτικών υπό τη συγκυρία μιας κρίσης πρέπει να επανεπισεργαστούμε αυτές τις πολιτικές και αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν ακούστηκε το όνομα. Η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Θέλετε να λάβετε εσεί τον λόγο, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαι επικεφαλής της μονάδας για πολιτική, την πολιτική για τους νέους. Με συνοδεύουν δύο συνάδελφοι, ο κύριος Γιώργεν Χάνσεν, επικεφαλής αρμόδιος για τον διαθρωμένο διάλογο και εκ δεξιών μου Φένστατ από την Νορβηγία, εθνικός επαίων, ο συντάκτης της έκθεσης για τις, για τους νέους στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του για το συνεχόμενο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό και το ζήλο της για την εμβάθυνση και τη διεύρυνση της στρατηγικής για τους νέους. Θυμάμαι και για από παλαιότερες ε, ε, στιγμές πόσο, με πόσο ενδιαφέρον στρέψατε την προσοχή σας σε αυτή τη στρατηγική και υποβάλατε προτάσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει διατομεακή ισχυρή έμφαση σε αυτή τη στρατηγική για τους νέους. Οκτώ άξονες στρατηγικής έχουμε από την απασχόληση, τον εθελοντισμό, τους νέους και τον κόσμο και είναι αρκετά πολύ ισχυρής. Ε, υπάρχει αρκετή πολυμορφία. Το σχέδιο το οποίο θα έχετε δει όλοι, ενημερωτικά το αναφέρω, βασίζεται στις εθνικές εκθέσεις όλων των επιμέρους κρατών μελών. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν είναι κάτι που έκανε μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μόνη της. Ενημερωτικά υπάρχει και το τμήμα για την επικοινωνία, 12 σελίδες περίπου επικοινωνία, που αφορά επικοινωνία από εμάς Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εμάς Ευρωκοινοβούλιο. Και τα δύο έγγραφα την προσέγγισή μας στη νέα πολιτική για τους νέους. 100 σελίδες το κάθε έγγραφο περίπου. Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και άλλα στοιχεία για τις τάσεις που ακολουθούνται και, σημειώνονται σήμερα για τους νέους. Είναι θλιβερό το ότι δυστυχώς το πεδίο πολιτικών για τους νέους δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη σημερινή μακροοικονομική κατάσταση. Είναι θλιβερό ότι η ανεργία των νέων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ουράνια, έχει εκραγεί και έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσφέρουμε λύσεις υπό τη μορφή ιδιαίτερα άτυπης μάθησης και εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε αυτό και προηγούμενα, επενδύοντας στις δεξιότητες, ατομικές δεξιότητες των νέων. Συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική στο νέο πολιτικό πεδίο, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να δώσουν feed-in, να συμμετάσχουν στις προτάσεις για την απασχόληση που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Γενική Διεύθυνση μέσω ενός διαρθρωμένου διαλόγου. Διαρθρωμένου διαλόγου όπου η απασχόληση των νέων είναι το θέμα του πρώτου κύκλου από το 2010 στα μέσα 2011. Το φόρουμ των νέων και μάλιστα κατά τη διάρκεια αυτής, αυτού του κύκλου και στον κύκλο συμμετοχής που ολοκληρώνει συμμετοχής που είναι κυρίαρχη προτεραιότητα μέσα στο πλαίσιο του διαφρομένου διαλόγου στον πρώτο αυτοκύκλο για τις, την πολιτική, της μας για τους νέους. Και πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό μέσο για τα κοινωνικά μέσα αυτά, αυτό. Ε, σημαντική προσέγγιση. Οι νέοι με δεδομένη αυτή την θέσπιση αυτού του πλαισίου εργαστήκαμε ώστε να υπάρξει μια μελέτη από το LSE London School of Economics για τη συμμετοχή που ε, σύντομα θα ε, δημοσιοποιηθεί. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για τα social media, για τα μέσα και για την συμμετοχή των νέων και πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτή. Προσδοκούμε ότι σύντομα θα μπορέσει να δημοσιευτεί. Βρίσκεται στο ε, καθοδόν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι διαθέσιμη αλλά α, ας το πω έτσι την επεξεργαζόμαστε για να αποκτήσει μια περισσότερο κοινωνική έκδοση στην φάση, ε, πρώτη φάση δημοσιοποίησης ε, στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσουμε έτσι μια νέα ε, φιλοδοξία να αρχίσουν τα νέα μέσα να ανοίγονται προς τους νέους και οι νέες τεχνολογίες και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους νέους. Αυτό για να ληφθεί και αυτό υπάρχει υπόψη τονίζοντάς το. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Υπάρχουν πολλά θέματα, πολύμορφα. Οι πολιτικές για του νέου είναι πολύ Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες και σε άλλους τομεί που προανέφερα. Η συμμετοχή των νέων και η Βόρεια Αφρική αναφέρθηκε. Ο ρόλος των νέων στις επαναστάσεις στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Θα ήθελα να πω ότι είχαμε και ένα μείζον γεγονός με το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Τίνιδα όπου είχαμε νέους ακτιβιστές και νέους ε, ε, ηγέτες των νέων παρόντες πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η πολιτική σε αυτή την περιοχή για τους νέους. Στέφθηκε με επιτυχία αυτό το εγχείρημα και αυτό έγινε πριν από τα πρόσφατα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική με την επίθεση κατά της ε, Αμερικανικής Πρεσβείας ε, στη Λιβύη και τα λοιπά και όλα τα συναφή. Ένα, ε, μια εκδήλωση πραγματικά υψηλότατου επίπεδου. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο ήταν πρωτοπόρο ε, ως πρωτοβουλία. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αυτή είναι μια σύντομη, συντομή απάντηση σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ. Ποιος από συναδέλφους θα ήθελε να λάβει τον λόγο, να παρέμβει. Από συναδέλφους σας κάποιος θέλει να παρέμβει. Θέλει να πει κάτι okay. Δεν συμβαίνει. Εντάξει λοιπόν. Ο κύριος Παπα-Νικολάου λοιπόν. Έχετε τον λόγο για να ολοκληρώσετε κύριε Παπα-Νικολάου. Very briefly. Ε, Εν συντομία ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδελφούς για τα σχόλιά τους και προσδοκώ να συνεργαστώ με τους Κιώδης. Ε, πιστεύω ότι θα είναι επικοδομητική και δημιουργική η ευκαιρία αυτή για όλους μας για να επαναλάβω κάτι ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Γνωρίζω τους συναδέλφους από την Κομισιόν, έχουμε συνεργαστεί στην αρχική έκθεση για τη στρατηγική για την νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι βέβαιος ότι θα ξανασυνεργαστούμε καλά και ήθελα να τους ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολλά και στην αρχική μας έκθεση χαιρετήσαμε όλες αυτές τις προσπάθειες και όλα τα νέα εργαλεία που εισάγουν στον τομέα των πολιτικών για την νεολαία. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο είμαι λιγότερο ενθουσιώδη, ίσως λίγο απογοητευμένος και απεσιόδοξος για ορισμένα ζητήματα, είναι ότι βρισκόμαστε εν μέσω μια τεράστια κρίση. Πιστεύω ότι δεν είμαστε επαρκώς αποτελεσματικοί. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη και δεν παρέχει την έμπνευση που θα θέλαμε. Και πιστεύω ότι σήμερα με τα νούμερα που έχουμε μπροστά μας δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους για τις στρατηγικές 2020. Και ε, φυσικά δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε διαδομιακή προσέγγιση στις λύσεις που προτείνουμε. Ανέφερα ορισμένα παραδείγματα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και φυσικά πιστεύω ότι στο πλαίσιο των συζητήσεών μας τις επόμενες εβδομάδες. Ε, ορισμένες από αυτές με τη συμβουλή της ε, Κομισιόν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην Επιτροπή μας, όχι γιατί θέλουμε να επικρίνουμε ή να είμαστε αρνητικοί όσον αφορά ορισμένα από τα συμπεράσματα, αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί και να συμπεριφερόμαστε με τρόπο που υποδηλώνει την επίγουσα ανάγκη και να δράσουμε αποτελεσματικά, αποφασιστικά σε αυτό το τομέα. Θεωρούμε ότι αποτελεί απειλή για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, μπορούμε να ολοκληρώσουμε έτσι το, το τελευταίο αυτό σημείο στην ημερησία διάταξη. Και περάμε στο σημείο 10, συνάντηση τώρα των συντονιστών, ε, έγκριση των απαντήσεων των αποφάσεων των συντονιστών. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Διάφορα, δεν υπάρχει τίποτα. Επόμενη συνεδρία 26-27 Νοεμβρίου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς και εύχομαι σε όλους σας καλό βράδυ. Γεια σας.